Ja, Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε τη συνεδρία που διακόπτει εχθές και σας καλωσορίζω εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Έχουμε προβλέψει για, την, ε, ε, για το πρωινό μας σήμερα μία δημόσια κρόαση για την ε, ενίσχυση της Ελλάδας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται. Είναι πολλοί οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα. Ελλάδα στην οποία έχει προβλεφθεί μια ειδική μορφή βοήθειας, η λεγόμενη Task Force, μια ομάδα που έχει ε, προβλεφθεί να προσφέρει τη βοήθειά της. Και έτσι σήμερα έχουμε εδώ τους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε το πώς μπορεί, θα μπορούσε να συνδράμει την Ελλάδα η Task Force. σε ποιο βαθμό γίνεται δεκτή ε, η βοήθειά της, ε, πώς αξιοποιείται πού μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα, τι μπορούμε να διδαχθούμε για το, για το μέλλον. Και αυτό στη γραμμή των όσων έχει και από τον κανονισμό και το περάρτημα 7 που ορίζει τα κύρια καθήκοντά της, επομιστεί η Επιτροπή Ελέγχου του, κανονισμού, του Προϋπολογισμού. Έχω λοιπόν εδώ μεγάλες προσωπικότητες, ειδικού προσκεκλημένους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχω καταρχάς τον κύριο Χόρστ Ράιχενμπαχ, τον επικεφαλής της ε, Task Force για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ, κύριε Ράιχενμπαχ. Επίσης, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω τον κύριο Στέφανο Μάνο, πρώην ε, Υπουργό των Οικονομικών στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Και στη συνέχεια θα, θα ακούσουμε και τον κύριο Νόρμον Σπόπενς, αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κύριο Πέτερ Στούπ Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θα έχουμε τον κύριο Μπεν Κνάπεν, Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον κύριο Wolf από το Think Tank. Μπρούχελ, που θα είναι παρόντες, θα συμμετάσχουν στη συζήτησή μας. Σας καλωσορίζω όλους και πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο Χατζημαρκάκη, τον συνάδελφο και εισηγητή, θα ήθελα να κάνω τα εξής εισαγωγικά σχόλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε εγκαίρως το ερώτημα εάν πρόκειται να χρειαστεί χρηματοδοτική βοήθεια. Και προέκυψε ότι τα ταμεία συνοχής και τα διευθυντικά ταμεία δεν απορροφώνται όπως πρέπει στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν διαρκή προβλήματα, κανείς δεν τα εντοπίζει, κανείς δεν τα αντιμετωπίζει και έτσι όταν έρθει η ώρα να εξεταστούν τα συγκεκριμένα αίτια αυτών των προβλημάτων διαπιστώνεται ότι είναι πολλαπλά, δεν είναι ζήτημα μόνο της συγχρηματοδότησης ή της διοικητικής ικανότητας, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται με τις δομές λήψης αποφάσεων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να πάρουμε σαφείς απαντήσεις για το γιατί η Ελλάς δεν μπόρεσε να απορροφήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ικανοποιητικά τα κονδύλια της ε, χρηματοδότησης και τι υπάρχουν ε, με παραδείγματι ανάγκες. Υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται επιδοτήσει, αλλά δεν απορροφούν τα κονδύλια. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι χρειάζονται στήριξη αλλά δεν μπορούν να απορροφήσουν τα σχετικά κονδύλια. Και γι' αυτό λοιπόν τίθεται το ζήτημα τη πρακτικής βοήθειας. πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα να πληρώσουμε, να μην πληρώσουμε. Αυτό δεν είναι το ερώτημα για την Ευρώπη μα στην πραγματικότητα, το να πληρώσουμε, να μην πληρώσουμε. Το ερώτημα για την Ευρώπη είναι το πώ θα μπορέσει να καταστεί η Ευρώπη μια δομή αηφόρος, μια δομή βιώσιμη και έτσι έρχεται και το πακέτο διάσωση και ο προβληματισμό σχετικό με την σταθεροποίηση τη νομισματική πολιτική που θα πρέπει να ενισχύει και να σταθεροποιεί την πραγματική οικονομία. Και εδώ θα πρέπει τα αρμόδια όργανα οι διοικητικέ αρχές, τα θεσμικά όργανα να συμβάλλουν και να δώσουν αποφασιστικές απαντήσεις για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματο εν τέλει, γιατί πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Διαφορετικά θα είχαμε εμεί εδώ θέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού να συζητούμε αυτά τα θέματα. Σα ευχαριστώ λοιπόν που είστε όλοι εδώ. Και αν μου επιτρέπετε τώρα, θα ήθελα να καλέσω τον εισηγητή μα να κάνει την εισήγησή του. Ε, Ω προ τα πρακτικά αισθήματα πρέπει να σα επισημάνω ότι χθε βρέθηκε μέσα στην αίθουσα ένα iPad, ένα tablet και αν κάποιο από εσά του συναδέλφου ή από του ε, λοιπού που ήταν παρόντε στην αίθουσα χθε. το έχασε, α απευθυνθεί στη γραμματεία για να μπορέσουμε και εμεί να συγκεντρωθούμε στη δουλειά μα. Ε, για να μην έχουμε λοιπόν διακοπέ, δεν θα γίνει διάλειμμα για καφέ, ούτε θα μπουν δεν θα μπει το προσωπικό για να προσφέρει τον καφέ μέσα στην αίθουσα. Μπορείτε όμως να βγείτε έξω όπως θέλει και να σερβιριστεί. Η ε, συνεδρία μεταδίδεται από το διαδίκτυο, η διερμηνία διατίθεται στις συνήθεις γλώσσες και το λόγο έχει ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ράιχνμπαχ που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Η συνεδρίαση αυτή είχε προγραμματιστεί με υποδιαφορετικό τίτλο πριν από κάποιους μήνες. Αναβλήθηκε για διάφορους λόγους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας υποδεχόμαστε εδώ σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ και ο Στέφανος Μάνος ανάμεσά μας. Το ερώτημα λοιπόν που μας απασχολεί σήμερα και εδώ έχουμε και μια σχετική παρουσίαση, δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε στις οθόνες σας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων δαπανώνται κατά τρόπο που μπορούμε να έχουμε ωφέλη από την επένδυσή μας και εάν φυσικά ο στόχος επιτυγχάνεται. Η παρουσίαση είναι στις οθόνες, ωραία βλέπετε. Αν δείτε λίγο την ε, δήλωση της αποστολής της ε, ομάδας ε, για την Ελλάδα, της Task Force για την Ελλάδα, λέει ότι η Task Force είναι ένας πόρος στη διάθεση των ελληνικών αρχών καθώς αναζητούν τον τρόπο να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και ευμερούσα Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από οικονομικές ευκαιρίες και κοινωνική ισότητα και εξυπηρετείται από μια αποτελεσματική διοίκηση με ισχυρό ε, ήθος δημόσιας διοίκησης. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Με τον κύριο Ράιχα Χεμπάχ το καλοκαίρι του 2011 ξεκινήσαμε με πολύ καλό πνεύμα και αυτό είναι ο λόγος ύπαρξης της Task Force Αν δούμε λίγο την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, η άποψή τη είναι ότι η Task Force θα πρέπει να εντοπίσει και να συντονίσει την τεχνική συνδρομή που χρειάζεται η Ελλάδα προκειμένου να τηρήσει τους όρους ε, του Προγράμματος Προσαρμογής Ευρωπαϊκής Ένωσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα και φυσικά επωφελείται και της βοήθειας των υπολείπων κρατών μελών. Αν δείτε λοιπόν ε, έναν από τους στόχους ε, της Ελλάδος, μια ευημερούσα Ελλάδα, ε, δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η ανεργία αυξάνεται ε, και σύν το χρόνο ακόμα και περισσότερο. Και φέτος βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ποσοστό ανεργίας 27,2%. Είναι στην πρώτη θέση με την, Ελλάδα, ε, με την Ισπανία σε ποσοστά ανεργίας. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι η μετανάστευση. Λόγω της ανεργίας των νέων, άνω των, του 60% των νέων είναι άνεργοι, ένα στους δύο ε, κάτι παραπάνω και αυτό φυσικά είναι ζωφερό για το μέλλον και αν φυσικά αφαιρέσουμε το μέλλον των νέων, ουσιαστικά αφαιρούμε το μέλλον μιας ολόκληρης χώρας. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάλτιν Σούρτς, είπε πρόσφατα σε ομιλία του στο Συμβούλιο ότι πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι μας ενδιαφέρουν ε, τουλάχιστον συστημικά όσο και οι τράπεζες. Και αυτό εκφράζει την άποψη όλου του Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος Άντορ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τις κοινωνικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφάτως είπε, μάλιστα την περασμένη εβδομάδα, ξεκίνησε μια ε, πρωτοβουλία για να αρθούν οι γραφειοκρατικοί φραγμοί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε αργότερα και αυτό υποτίθεται ότι είναι μέσα στα καθήκοντα της Task Force. Από ό,τι φαίνεται σε κάποιους τομείς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα δεν λαμβάνουν αντίστοιχες επιστροφές από αυτά που επενδύουν ε, μέσω της ε, Task Force. Υπάρχει λοιπόν ένα ε, με πολύ μεγάλο ποσοστό μετανάστευσης ε, νέων Ελλήνων επαγγελματιών ε, με πολύ ψηλά προσόντα, ενώ ταυτόχρονα η Task Force για την Ελλάδα προσπαθεί να δώσει μια νέα όθηση στην απασχόληση μέσω περίοδων άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Από ό,τι γνωρίζω εγώ από τη Γερμανία, τη χώρα που γνωρίζουμε λίγο καλύτερα, η απασχόληση των νέων αυξήθηκε κατά 43% σε σχέση με το 2011. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν είναι εντυπωσιακά. Και πραγματικά νιώθω ότι βρίσκομαι και πάλι στην ε, δεκαετία του 60 όταν ο πατέρα μου αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα για να πάει στη Γερμανία να δουλέψει και η κατάσταση είναι αντίστοιχη σήμερα. Αν δούμε τώρα τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που θα δημιουργήσει ανάπτυξη απορροφώντα ευρωπαϊκά κονδύλια, διαπιστώνουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων έλαβαν μια κάποια μορφή ε, συνδρομή από την, τα όσα κάνει η Task Force στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο προβάλλεται είναι ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια και αυτό φυσικά είναι και το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Ε, προγράμματα σχεδιασμού, συντονιστικέ δραστηριότητε, ανταλλαγή ε, δεξιοτήτων ε, και γνώσεων. Είναι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εφαρμόζουμε και αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Κοινωνική ισότητα, που είναι και αυτός ένας από τους στόχους της αποστολής της Task Force. Τρία εκατομμύρια Ελλήνων ζουν στα όρια της φτώχειας. Τρία εκατομμύρια Ελλήνων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός. 500.000 παιδιά δίνουν μάχη για να επιβιώσουν σε οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να τους παρέχουν ούτε τα βασικά. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δύο χρόνια μετά την έναρξη της Task Force στην Ελλάδα, κύριε Ράχενμπαρκ, η Ελλάδα βιώνει κοινωνική κρίση και αυτή δεν είναι επίκριση προς εσάς, απλώς θέλω να το συζητήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να το υπερκεράσουμε αυτό. Πού ε, είναι τα εμπόδια και πού μπορούν να σταματήσουν αυτά τα ε, επονίδιστα στοιχεία που λαμβάνουμε κάποιοι εμπειρογνώμονε από άλλα κράτη-μέλη, ξέρω ότι έχουμε Γάλλου, Γερμανού, Ολλανδού συναδέλφου που ασχολούνται με θέματα αυτά, κάνουν ε, σύντομε επισκέψει για να ανταλλάξουν ε, ε, τεχνογνωσία και γνώσεις ε, με τους Έλληνες συναδέλφους. Αυτό από ό,τι φαίνεται όμως δεν αρκεί. Έχουμε μεγάλα προβλήματα επίσης στον τομέα της υγείας, που είναι ένας τομέας στον οποίο καλύπτεται και εσείς. Χιλιάδες ασθενείς ε, δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους. Ε, δεν υπάρχει δυνατότητα από τα νοσοκομεία να παρέχουν θεραπεία. Και έχουμε και ένα από τα πιο επωνύμιθα στοιχεία. Τα ποσοστά αυτοκτονιών έχουν φτάσει σε ποσοστά ρεκόρ τα επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα αναφέρονται σε, διπλασιαστό, ε, σε διπλασιασμό συγγνώμη, σε ένα χρόνο. Ε, υπάρχει μία αυτοκτονία την ημέρα. Δεν είναι καλό στοιχείο αυτό. Ε, στο παρελθόν υπήρχε συγγνώμη μία την ημέρα, τώρα είμαστε στις δύο αυτοκτονίες την ημέρα και αυτό ήταν το υψηλότερο ποσοστό τα τελευταία τρία χρόνια. Παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν θα επισέλθω πολύ στο θέμα της φοροδιαφυγής, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι αλληλένδετο με την κοινωνική ισότητα και φυσικά έχει και μεγάλη σχέση με το ερώτημα που τίθεται, γιατί οι φτωχοί είναι αυτοί οι οποίοι υπεβαρύνονται περισσότερο στην Ελλάδα. Ε, φορολογούνται οι πλούσιοι, δεν είναι κάτι βέβαια αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί σήμερα μας αποσχολεί η εφαρμογή της χρηματοοικονομικής βοήθειας, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι ο πλούτος που δημιουργείται στην Ελλάδα δημιουργεί ε, πρόβλημα και υπάρχει, ε, υπάρχουν φορολογικά εισοδήματα που στην Ελλάδα προέρχονται κυρίως από τους φτωχούς και όχι τόσο από τους πλουσίους. Φαίνεται ότι η κατάσταση για τους φτωχούς είναι ακόμα δύσκολη στην Ελλάδα. Θα ήθελα τώρα να σταθώ σε μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή, πολύ πιο σημαντική από τη φοροδιαφυγή και έχει σχέση με την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής βοήθειας, η διοικητική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς της αλλαγής στην Ελλάδα προκειμένου να φτάσουν τα λεφτά στην οικονομία, να φτάσουν τα χρήματα στη ε, προγράμματα. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στην Ελλάδα είναι ότι τα πάντα περνούν από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα, οποιαδήποτε απόφαση. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα στην Ευρώπη. Υπάρχει η Ισπανία, για παράδειγμα, η οποία ε, άλλαξε το σύστημά της. Υπάρχει η Γερμανία, η οποία είναι ομόσπονδο και έχει ε, άμεση ευθύνη για τα κρατήδια, για τα lender και στην Ελλάδα υπήρχε η μεταρρύθμιση Καλλικράτης που έκανε μία απόπειρα να απορρεφούνται τα κονδύλια απευθεία από τις περιφέρειες και οι περιφέρειες ε, και οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να συμμετέχουν περισσότερο ε, στην όλη διαδικασία. Διαπιστώνουμε όμως ότι ακόμα ευνοούνται οι πόλεις ε, ενώ η περιφέρεια της Ελλάδος αγνοείται. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Ράιχνμπαχ ε, το 2011, συγγνώμη, το 2012 εδώ στις Βρυξέλλες. Ήρθαν όλοι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες από την Ελλάδα να σας συναντήσουν και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας μεταξύ της Task Force και των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς από τις πληροφορίες μας ε, η επικοινωνία αυτή δεν φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ αυξημένα επίπεδα. Το ερώτημά μου είναι πόσοι ε, από τους προσώπους της Task Force εργάζονται απευθείας ε, στις περιφέρειες για να έχουν αυτή την άμεση επικοινωνία ε, η οποία θα πρέπει να γίνεται και καλύτερα. Πόσους ανθρώπους λοιπόν έχετε τοποθετήσει στις περιφέρειες ώστε να ασχολούνται άμεσα με τα στοιχεία αυτά. Διότι από τα στοιχεία που διαθέτουμε εμείς και μας στείλατε βέβαια και τα στοιχεία και απαντήσατε εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ερωτήσεις ε, που σας απευθύναμε για το πόσα ε, επενδύονται τα χρήματα τα οποία σας δίνουμε. Ε, έχουμε τα στοιχεία για το 2011 και για το 2012. Το 2012 ήταν και ένα πλήρες έτος και από ό,τι φαίνεται 840.138 ευρώ ε, έχουν δοθεί για το 2013. Δεν φαίνονται να είναι και πολλά αυτά τα χρήματα, αλλά το ερώτημα είναι ε, τι αποκομίζουμε εμείς από όλα αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας, ε, βέβαια, κύριε Ράιχνμπαχ, και να επισημάνω στο τέλος, διότι εγώ απλώς μια σύντομη εισαγωγή κάνω ως εισηγητής. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα σας κάνουν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις στη συνέχεια. Έχω ένα αριθματολόγιο, λοιπόν, το οποίο έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αρκετά λοιπόν ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρώτησα κατά πόσον αντιλαμβάνονται τι όσα κάνει η Task Force στην Ελλάδα ε, και κατά πόσον έχουμε μετριάσει τις συνέπειες της λιτότητας για τους Έλληνες, διότι τμήμα της πρότασης που έγινε ευθύς εξ αρχής όταν ξεκινήσατε το έργο σας ήταν να προσπαθήσετε να μετριάσετε τις επιπτώσεις της λιτότητας ε, που επιβάλλει η Τρόικα. Και ε, ζήτησα να υποβληθούν ερωτήσεις, λες και θα ήταν παρούντες ε, αυτοί που υποβάλλουν τις ερωτήσεις εδώ στη συνεδρίαση και αυτό το οποίο προέκυψε περισσότερο είναι γιατί η Task Force για την Ελλάδα δεν μετρίασε τις συνέπειες της λιτότητας ώστε να τις αντιληφθούν και οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβάνονται και πάρα πολλά από τα όσα κάνει η Task Force. Τι μπορούν να περιμένουν λοιπόν για το μέλλον. Εδώ έχετε το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου. Θεωρείτε ότι το έργο της Task Force ήταν επιτυχές κατά τρόπο που να το αντιλαμβάνεστε. Και από ό,τι βλέπετε η πλειονότητα λέει όχι. Εκρεμεί λοιπόν το ερώτημα πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, διότι αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό στοιχείο. Πρόκειται για κάτι το οποίο κάναμε μέσα σε τρεις μέρες. Ε, από το Σάββατο μέχρι τη Δευτέρα ρωτήσαμε ε, στα κοινωνικά ε, δίκτυα και συμμετείχαν περίπου 500 άτομα. Αλλά από ό,τι βλέπετε η άμεση απάντηση, η άμεση εικόνα που δίνεται είναι μάλλον αρνητική. Και αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κόσμος το έργο της Task Force. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να βελτιωθούμε διότι εδώ στα συμπεράσματα βλέπετε ότι παρά την παρουσία της Task Force, οι συνθήκες ε, στην καθημερινή ζωή στην Ελλάδα επιδεινώνονται συνεχώς παρά το γεγονό ότι η εικόνα ε, προ την Ευρώπη είναι καλύτερη, η αποτελεσματικότητα ε, τη χρήση των ευρωπαϊκών μέσων είναι αμφισβητήσιμη, δεν υπάρχει μια σαφή δομή, είναι αδιευκρίνιστος ο αριθμό του προσωπικού, παρά το γεγονό ότι στην απάντησή σα εσεί διευκρινίσατε πόσοι είναι, αλλά δεν ξέρουμε πόσε είναι οι διμερεί επαφέ και από εκεί και πέρα ε, τα αποτελέσματα δεν γίνονται αντιληπτά ικανοποιητικά. Θεωρούμε λοιπόν ότι η Task Force θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ε, καθημερινή ζωή των ανθρώπων, θα πρέπει να γεμφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, να υποστηρίξουμε την περιφέρεια και όχι τις μεγάλες αστικές περιοχές, να υπάρχει μια σαφέστερη δομή και συγκεκριμένο προσωπικό και θα πρέπει να προσμετράτε και αποτελεσματικότητα ώστε να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ κύριε Ράιχενμπαχ που είστε εδώ σήμερα στην ακρόαση. Thank Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χατζημαρκάκη, γιατί πραγματικά έθεσε σειρά ερωτήσεων. Δείχνει την δέσμευσή του. Πληθώρα πληροφοριών ε, μας έδωσε ο κύριος Χατζημαρχάκης. Και τώρα θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες, αυτούς που πραγματικά έχουν αναλάβει αυτήν την αποστολή που συνοδεύουν με την ε, γνώση τους αυτήν την επιχείρηση στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε καταρχήν τον Horst Reichenbach. 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, λίγο πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα αναγκαστώ να εγκαταλείψω την Προεδρία. Ο Αντιπρόεδρος θα με αντικαταστήσει για περίπου μία ώρα. Κύριε Ράχενμπαχ, έχετε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που θα μας κάνατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν που με προσκαλέσατε εδώ μετά από 20 μήνες αποστολής της Task Force, της ομάδας δράσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε εδώ με την Επιτροπή σας πώς έχει διεκπαιρεώσει μέχρι τώρα η ομάδα δράσης την αποστολή της στην Ελλάδα και είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας παρουσιάσω τα θέματα αυτά. Καταρχήν άκουσα τον εισηγητή, ο οποίος έδωσε διάφορες ενδείξεις, διάφορα στοιχεία της εντολής της ομάδας δράσης, η οποία βεβαίως ε, ουσιαστικά τον Σεπτέμβριο 2011 ξεκίνησε δύο συστατικά, αν θέλετε, αποτελούν αυτή την εντολή, συντονισμός της τεχνικής βοήθειας, την οποία χρειάζεται η Ελλάδα για να μπορέσει πραγματικά να ε, διεκπαιρεώσει το πρόγραμμα προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε τεχνική βοήθεια, να στηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτό το έργο. Και δεύτερον, σύσταση νομοθετικής, κανονιστικής, διοικητικής και ενδεχομένως ανασχεδιασμός μεταρρύθμισης έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να απορροφήσει με καλύτερο και πιο γρήγορο τρόπο τα διαρθρωτικά ταμεία, τα κονδύλια που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Θα ακολουθήσει μία παρουσίαση με πολλά στοιχεία, πολλά, πολλές λεπτομέρειες θα έλεγα. Έχετε όλα αυτά εξάλλου ε, στην γραπτή μου παρουσίαση, στο PowerPoint. Εγώ θα επικεντρωθώ σε κάποια σημεία που τα θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα οποία θα πρέπει εδώ να σας παρουσιάσω, ιδιαίτερα τα οικονομικά στοιχεία, γιατί πιστεύω ότι είναι εξάλλου και η ιδιαίτερη αδομοδιότητα της Επιτροπής σας. Θα σας δώσω και μία γενική εικόνα των διαφόρων τομέων στους οποίους εμπλέκεται η ομάδα δράσης. Καταρχήν επιτάχυνση πολιτικής συνοχής, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βλέπετε μία σειρά από άλλες δραστηριότητες τρεις σημαντικοί τομείς στους οποίους εντοπίζουμε την εργασία μας σαν ομάδα δράσης μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς και άλλα κράτη-μέλη, προϋπολογισμός, φορολογία, μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικό περιβάλλον πρόκειται για τομείς στους οποίους οι διαρθρωτικές αδυναμίες και ελλείψεις της Ελλάδας είναι σημαντικές και σε αυτούς εμείς εντοπίσαμε τις προσπάθειές μας. Τώρα, με ποιο τρόπο εκτελούμε την αποστολή μας στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω ότι συνεργαζόμαστε πολύ στενά με άλλα κρατημέλη, με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς αλλά θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση εδώ στο σημείο εκκίνησης όλων των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Αυτό το κάνουμε μετά από αίτηση των ελληνικών αρχών. Πρόκειται για μια εντολή που μας έχει δοθεί από τις ελληνικές αρχές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ουσιαστικό θα έλεγα για την αποτελεσματικότητα της ε, εργασίας αυτής της ομάδας δράσης. Και εδώ έχουμε διάφορα παραδείγματα τομέων στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και είναι ενδεικτικοί. Είμαστε παρόντες σε πάνω από 100 προγράμματα και σχέδια στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά την μέθοδο εργασίας μας, θα έλεγα ότι ο πρώτος τρόπος παρέμβασης είναι μία διερεύνηση, ένας εντοπισμός από κοινού με τις ελληνικές αρχές για το ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες που μπορούμε εμείς ε, να εντοπίσουμε και να διερευνήσουμε αδυναμίες. Αυτό μας, ε, ε, σε αυτό μας καθοδηγεί βεβαίως η εντολή της Τρόικας. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Και αυτό έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό αν θέλετε, με σχέδια δράσης, ε, χάρτες πορείας και οι περισσότεροι τομείς τους οποίους σας περιέγραψα έχουμε ενεργοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε εντοπίσει πολύ συγκεκριμένα από με τις ελληνικές αρχές ποιοι είναι οι τομείς τους οποίους θα πρέπει να παρέχουμε την τεχνική μας βοήθεια. Αποστολές λοιπόν εμπειρογνωμόνων εργαστήρια, διερευνητικές αποστολές οργανώθηκαν στην Ελλάδα. Βλέπετε εδώ ουσιαστικά ότι πρόκειται για πολλές αποστολές, τις οποίες συμμετέχουν πάνω από 20 κράτη-μέλη. Η ομάδα δράσης συντονίζει κατά κάποιο τρόπο στις ε, συναντήσεις που οργανώνει με όλα αυτά τα κράτη-μέλη και με τους άλλους διεθνείς οργανισμούς την αποστολή μας στην Ελλάδα. Βλέπετε εδώ τις πιο δραστήριες χώρες που παρέχουν τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βεβαίως και συμβούλους εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχουν ε, και συμβάσεις με εταιρείε συμβούλων ιδιωτικές για την παροχή βοήθειας και βεβαίως από τη στιγμή που δεν αρκεί αυτή η βραχυπρόθεσμη παροχή εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης, βλέπετε εδώ την οικονομική πλευρά αυτής της βοήθειας, της συμβάσεις 850.000 ευρώ. Είναι το συνολικό ποσό αυτών των συμβάσεων ε, των εμπειρογνωμόνων που χρηματοδοτούνται βεβαίως από τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρεις τομείς. Βλέπετε τα έσοδα. Και βεβαίως βλέπετε και τους τομείς, ε, τη διοικητική μεταρρύθμιση, το επιχειρηματικό περιβάλλον, στους οποίους ε, είμαστε ενεργοί μέχρι τώρα. Πρόκειται για κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναλαμβάνω, για μια σειρά φορέων, διεθνών και εθνικών. Επίσης θα ήθελα να επαναλάβω εδώ ότι η ομάδα δράσης δεν έχει δική της χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τα κοινωνικό ταμεία, τα περιφερειακό ταμεία και η διαχείριση γίνεται όλων αυτών των κονδυλίων από έναν αρμόδιο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Και ο Πίτερ Γιόργενσεν θα σας κάνει μια παρουσίαση αυτού του τμήματος της αποστολής μας. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι έχουμε συνάψει συμβάσεις, ότι τα κονδύλια προέρχονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και ότι πραγματικά στοχεύουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που παρέχουν μια συγκεκριμένη εμπειρία, τεχνογνωσία Οι αποστολές του ΩΣΑ χρηματοδοτούνται από ελληνικές πηγές. με σκοπό την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Στην επόμενη διαφάνεια μπορείτε να δείτε, όπως σας είπα, την προέλευση των πόρων. Όσον αφορά την προετοιμασία ιδιαίτερα των δράσεών μας για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών αλλά και της διοικητικής ε, μεταρρύθμισης, κάτι που προϋποθέτει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι απτό στον οικονομικό τομέα. Τα αποτέλεσματα αυτά σαφώς ε, θα είναι πρόθεσμα Σήμερα, μετά από πέντε χρόνια ύφεση, η ανεργία στην Ελλάδα είναι σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και έχουν ξεκινήσει κάποιες ε, δράσεις, κάποιες δραστηριότητες για την βελτίωση αυτών των τομέων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε, όπως είπε και ο πρόεδρος στα εισαγωγικά του σχόλια, υπάρχει σημαντική ανάγκη για ρευστότητα η οποία θα τροφοδοτήσει την πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει εδώ με διάφορους ε, φορείς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ταμείο Επενδύσεων, και το ΕΤΕΑΝ την βάση για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Και βλέπετε εδώ ότι 2,6 δις είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι περίπου το 1%, πάνω από το 1% του ελληνικού ΑΕΠ. Βλέπετε επίσης ότι οι πραγματικές πληρωμές μέχρι τώρα από αυτό το ποσό είναι εξαιρετικά λίγες. Προσπαθούμε λοιπόν από κοινού με το μηχανισμό σταθερότητας αλλά και με τις τράπεζες να βελτιώσουμε την ε, τροφοδοσία της ελληνικής οικονομίας και την καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Εδώ βλέπετε την ροή των κονδυλίων και πάλι βλέπουμε την ίδια εικόνα. Απλώς εδώ η, ο πίνακας αυτός σας παρουσιάζει τους αριθμούς με διαφορετικό τρόπο. Τα δάνεια που έχουν δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω κάποια παραδείγματα πριν ολοκληρώσω της τεχνικής βοήθειας που παρέχουμε στην Ελλάδα και η οποία έχει ήδη ε, αποτελέσματα. Όσον αφορά την διοικητική μεταρρύθμιση, την κεντρική ε, διοίκηση, είναι μία από τις προτεραιότητες από κάθε πλευρά. Περισσότερα, τα περισσότερα ελληνικά υπουργεία έχουν περάσει από μία διαδικασία αξιολόγησης. Πάνω από 206.000 άτομα εργάζονται στον τομέα αυτό και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για την μείωση των δημόσιων υπαλλήλων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αυτήν την ε, μεταρρύθμιση ακολουθώντας την σύσταση της έκθεσης του ΟΣΑ θεσπίζοντας ένα Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την οποία στηρίζει η ομάδα δράσης. Μια άλλη πάρα πολύ σημαντική επιχείρηση στην Ελλάδα είναι οι παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων, κάτι που έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται η ομάδα και οι ελληνικές αρχές τους τελευταίους 20 μήνες. Τα ωφέλη από το ξεκίνημα αυτών των έργων, την επανεκκίνηση θα έλεγα αυτών των έργων, θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για το ελληνικό ΑΕΠ και είμαστε στην τελευταία φάση της διευθέτησης έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν εκ νέου τα έργα. Κάτι που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, μετά από πολλούς μήνες αβεβαιότητας για αυτά τα πολύ σημαντικά έργα υποδομής, ελπίζουμε το Ελληνικό Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να δώσει το πράσινο φως για να ξεκινήσουν εκ νέου αυτά τα έργα. Όσον αφορά τη διευκόλυνση των εξαγωγών, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη διαδικασία με σκοπό να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος κατά 50%, να αυξηθούν κατά 10% οι εξαγωγές από την Ελλάδα, κάτι που θα έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και πολύ συγκεκριμένα η αξιολόγηση δύο πολύ σημαντικών ελέγχων στις προτελωνιακές διαδικασίες έχει ολοκληρωθεί. Και θα ήθελα να σας δώσω και ένα τέταρτο παράδειγμα αποτελεσματικής δράσης που είναι η μεσολάβηση σε υποθέσεις που χρονοτριβούν, που πολλές φορές ε, παίρνουν πάνω από πέντε χρόνια στην Ελλάδα για να διεκπεριωθούν από τις δικαστικές αρχές. Πρόκειται λοιπόν για την ε, δυνατότητα εξοδικαστικής διευθέτησης κάποιων υποθέσεων και η ομάδα δράσης έχει συμβάλει στην κατάρτιση των ε, μεσολαβητών με αυτό τον τρόπο συνεισφέρουμε παρέχοντας στοιχεία πληροφορίες, κάτι που ξεκίνησε πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα. Ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο δεν είναι στην διαφάνεια που βλέπετε, είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς. Υιοθετήθηκε ένας νόμος πρόσφατα στην Ελλάδα για την καταπολέμηση της διαφθοράς με πιο συστηματικό τρόπο. Έχει οριστεί ένας συντονιστής αρμόδιος για τα θέματα αυτά, κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα την διεκπαιρέωση αυτής της αποστολής. πολέμηση λοιπόν της διαφθοράς στην Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι βεβαίως ε, η τεχνική βοήθεια που προσφέρουμε ενεργοποιείται σε διάφορους τομείς σημαντικούς πολλοί Ξεκινούμε από την ανάλυση, τη διερεύνηση μέχρι την υλοποίηση. Και βεβαίως αυτό είναι λογικό να έχει πάρει κάποιο χρόνο. Εδώ και 20 μήνες εργαζόμαστε για την διεκπαιρέωση αυτής της αποστολής. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει λιγότερο από ένα χρόνο στην εξουσία η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και την ομάδα δράσης και τα διάφορα κράτη-μέλη και διεθνείς οργανισμούς προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι τα μέσα του 2015 και όσον αφορά αυτήν την ε, τεχνική βοήθεια που παρέχουμε και την αποτελεσματικότητά της, αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την όθηση που θα δώσουν οι ελληνικές αρχές σε αυτήν την διοικητική μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Ράχινμπαχ για την παρουσίαση. Μας έχουν ζητήσει το λόγο ορισμένοι συνάδελφοι. Θα προτείνω λοιπόν οργανωτικά να προβλέψουμε στις 11 την συζήτηση, γιατί έχουμε ήδη μια καθυστέρηση σημειώσει. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Στέφανο Μάνο, πρώην Υπουργό των Οικονομικών. Το παρακαλώ να λάβει το λόγο. Είναι γνωστό ιδιαίτερο διότι τα τελευταία 20 χρόνια ήταν εκείνο ο οποίο έκρουε τον κόδωνα του, του κινδύνου για τι υπερβολικέ δαπάνε και το χρέο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ και κύριε Μάνο, σα δίνω το λόγο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ που με δέχεστε εδώ να μιλήσω. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Θα προσπαθήσω, ξεκινώντας, να κάνω μια επισκόπηση της κατάστασης στην Ελλάδα όπως εγώ τη βλέπω. Μια επισκόπηση με την οποία θα ήθελα και να υπογραμμίσω ορισμένες παρατηρήσεις για το έργο της ομάδας δράσης, της Task Force. Πριν ξεκινήσω ωστόσο, θα ήθελα να απευθύνω ένα ευχαριστώ στον κύριο Ράχενμπαχ για την ε, ενσυναίσθηση προς την Ελλάδα και την, ε, το αίσθημα ενσυναίσθησης με το οποίο συνεχίζει το έργο του για την Ελλάδα. Η δημοσιονομική προσαρμογή και η πρόοδος αυτή ήταν εντυπωσιακή οι δαπάνες εκτός στόχων το 2009 ήταν 112, 113 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Συνολικές δαπάνες λοιπόν το 2009, ενώ εφέτος αναμένεται να πέσουν στα 79 δισεκατομμύρια. Τέσσερα χρόνια με 30% μείωση μέσα στα 4-7 χρόνια στις δαπάνες, στις κρατικές, ένα πολύ εντυπωσιακό επίτευγμα. Η προσαρμογή αυτή λοιπόν κατέστη δυνατή χάρη σε σημαντικές περικοπές σε μισθούς και κοινωνικές παροχές από ένα αρνητικό πρωτογενές, από ένα πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού σε ύψος 24 δισεκατομμυρίων το 2009, αναμένεται τώρα το 2013 μηδενικό έλλειμμα, ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Μπορεί, μέσα σε τέσσερα χρόνια δηλαδή μπορέσαμε να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Το επίτευγμα όμως αυτό είχε τεράστιες παράπλευρες απώλειες, τεράστιο παράπλευρο κόστος, κόστος στο λαό, διότι έγινε αυτή η δημοσιονομική προσαρμογή με συνέπεια την συρρήκνωση κατά 25% της οικονομίας, τον τριπλασιασμό του αριθμού των ανέργων κατά 27%, στο 27% και ιδιαίτερος, χαρακτηριστικό είναι το φαινόμενο της επιδημικής ανεργίας των νέων σε ύψος 65% τελευταία νούμερα στα, στη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία, έχουμε 74% τελευταία στατιστικά στοιχεία νέοι χωρίς δουλειά. Πρόκειται για μια επιδημία ανεργίας. Λόγω της συρρήκνωσης λοιπόν και της απότομης ραγδαίας αύξησης της ανεργίας, άρα άνεργοι οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν τους φόρους τους, έγινε αναγκαία επίση η ραγδαία αύξηση των φόρων, ώστε να πληρώνουν περισσότερους φόρους αυτοί που ακόμη έχουν δουλειά. Άρα έχουμε κόσμο χωρίς δουλειά και αυτοί που έχουν μια θέση εργασία καλούνται να πληρώσουν ακόμη περισσότερους, πολύ περισσότερους φόρους από ό,τι πριν, προκειμένου να καλύψουν το έλλειμμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι περιθώριο για άλλες αυξήσεις φόρων ή για περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων δεν υπάρχει κατά με. Ο κίνδυνος μάλιστα είναι, κατά να αντιστραφεί απότομα αυτή η δημοσιονομική λιτότητα, η πολιτική της λιτότητας, όταν δηλαδή καταστεί ανυπόφορο πλέον, ανυπόφορος αυτός ο φόρτος, αυτή η πίεση για το λαό. Υπάρχει ο κίνδυνος να αναστραφούν πλέον, να αλλάξει πορεία και η κυβέρνηση ακόμα εφόσον αυτό καταστεί πολιτικά ανυπόφορο για το λαό. Θα σας εξηγήσω το πρόβλημα πώς το βλέπω. Το πρόβλημα για μένα ήταν και είναι η απουσία βούλησης από πλευράς της, ε, του ελληνικού πολιτικού συστήματος για εισαγωγή βαθέων μεταρρυθμίσεων ε, διαρθρωτικών που θα αντιμετώπιζαν τη φοροδιαφυγή και θα απελευθέρωναν και θα καθιστούσαν πιο ευέλικτη την αγορά εργασίας. Ιδιαίτερα δε η ιερή Αγελάδα είναι το δημόσιο. Η ιερή Αγελάδα που δεν τολμά κανείς να την αγγίξει είναι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα και καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να την αγγίξει ε, πειράξει. Αυτό οδηγεί σε μία απολύτως δυσλειτουργική γραφειοκρατία. Μέσα στο πλαίσιο αυτό καλείται η ομάδα δράσης να προσφέρει, να επιτελέσει το έργο της, την εντολή της, που είναι εισαγωγή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι βλέπω εγώ το έργο της ομάδας δράσεως, να βοηθήσει δηλαδή στην εισαγωγή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα κληθεί να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Το τι θα γίνει με τη δημόσια διοίκηση, το τι θα γίνει με το νομοθετικό πλαίσιο και τους θεσμούς που, θα προωθήσουν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Αυτή θα ήταν η δουλειά, αυτή είναι η δουλειά της ομάδας δράσης, ή ασδήποτε ομάδας δράσης. Και έχουμε τώρα την ε, τριμηνία έκθεση του κυρίου Ράχενμπαχ που μας δείχνει ε, το εύρος και πλάτος και βάθος των προσπαθειών για παροχή βοήθειας στην Ελλάδα. Είδατε ότι πρόκειται για εκατοντάδες έργα και σχέδια. Μεγάλη προσπάθεια λοιπόν. Πλην όμω η αποτελεσματικότητα της ομάδας δράσης εξαρτάται από την βούληση του προσών συνδρομή, δηλαδή της Ελλάδας να δεχθεί τη συνδρομή αυτή. Ό,τι συνδρομή και να προσφέρουμε, ό,τι αρρωγή και να προσφέρουμε, εάν ο προσόν δεν θέλει να τη δεχθεί, τότε δεν έρχεται κανένα αποτέλεσμα. Στη δε δική μας περίπτωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν βλέπω εκδήλωση τέτοιου είδου βουλήσεως για αποδοχή της αρρωγή. Τουναντίον αντίον βλέπουμε παντού προσκόμματα και εμπόδια, διότι κανείς δεν τολμάει να αγγίξει, να ακουμπήσει την Ιερή Αγελάδα. Θα χρειαστήσω να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να επιτύχει ουσιαστική και μακροπρόθεσμη διοικητική μεταρρύθμιση χωρίς μια απότομη ρήξη και επανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό απαιτεί λοιπόν ριζική περικοπή του αριθμού των μη ε, ικανών των περιττών υπαλλήλων. Είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα, είναι πολλοί οι οποίοι περιτεύουν, περισσεύουν και θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία συγκεκριμένα ε, είχα εκτιμήσει δηλαδή πριν από μερικά χρόνια ότι πάνω από 400.000 εργαζομένων από το 1,5 εκατομμύριο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα θα έπρεπε σε περίοδο 4-5 ετών να αποχωρήσουν. Η Τρόικα έκανε μια προσπάθεια για να πιέσει προς το στόχο της απόλυση 150.000 έως το 2015. Τώρα ε, αναλογίστε τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί ε, έστω και για 15.000. Εγώ λέω 400.000, η Τρόικα μέχρι 15 για αυτές τις 15.000 που είναι μεγάλο θέμα συζήτησης, αυτές τις 15.000 λοιπόν περιλαμβάνουν ε, απατεώνες, ε, ψυχασθενείς και διάφορους άλλους οι οποίοι παραμένουν στα έστους και παίρνουν μισθό. Δεν έχει ακόμη δώσει αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση μεταξύ της Τρόικα και της κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να δώσει αποτέλεσμα ουσιαστικό, δυστυχώς. Και θα ήθελα να σας πω ότι από ό,τι έχω ακούσει στην Ινδία δεν επιτρέπεται μία αγελάδα η οποία ακόμη και αν αφοδεύει στη μέση του δρόμου και ενοχλεί, δεν μπορεί να την ακουμπήσει κανείς, δεν μπορεί να την μετακινήσει κανείς και μένει στη μέση του δρόμου να αφοδεύει. Αυτό λοιπόν θα έλεγα είναι ο παραλληλισμός με την αντιμετώπιση την οποία επιφυλάσσουμε στους υπαλλήλου του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, γιατί κανείς δεν αξιολογείται, κανείς δεν υφίσταται ε, μομφή ή κυρώσεις, κανείς δεν παίρνει συγχαρητήρια ή έπαινο για τις καλές του επιδόσεις και κανείς δεν απολύεται. Και έτσι φτάνουμε στο ζήτημα που έθιξε και ο κύριος Ράχενμπαχ, που είναι το βαθύ, η βαθιά ανάγκη για μεταρρύθμιση και της του φορολογικού συστήματο. Βεβαίω και χρειάζεται αυτό. Βεβαίω χρειάζεται μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο, αλλά δεν πρόκειται να γίνει μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματο όσο παραμένουν στο απειρόβλητο όσοι δουλεύουν στι εφορίε. Πάλι μέσα στο σύνδρομο αυτό τη Ιερή Αγελάδα. Και επίση θα πρέπει να σα επισημάνω ότι το σύστημα αυτό το φορολογικό είναι κομμάτι του γενικότερου διοικητικού συστήματο. Δεν μπορεί δηλαδή να αποκοπεί και να εξεταστεί χωριστά. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξάγει περισσότερο, θα πρέπει να παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά ως προς τα εισαγόμενα. Βεβαίως έχει παρουσιαστεί μια βελτίωση στο ισοζύγιο ε, το εμπορικό το τελευταίο διάστημα, καθώς είναι αναγκασμένες οι επιχειρήσεις πολύ συχνά να εξάγουν και κάτω από το κόστος προκειμένου να διατηρήσουν την ε, ικανότητά τους την παραγωγική. Χρειάζεται δηλαδή η ρευστότητα και προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτό για να μην κλείσουν ε, εξάγουν ακόμη και κάτω από το κόστος. Ε, μία όμως ε, ουσιαστική ανάπτυξη των εξαγωγών θα απαιτεί πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει η μείωση των μισθών. Πολύ περισσότερα πράγματα χρειάζεται για να βελτιωθούν οι συνθήκες και να έχουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται απλούστευση, απλούστευση του φορολογικού συστήματο, του νομοθετικού πλέγματος, τις ε, ιδιωτικοποιήσεις ε, χρειάζεται να ε, ελαφρυνθεί αυτή η γραφειοκρατική επιβάρυνση η οποία δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Και θα είμαι πολύ ειλικρινής δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη στην Ελλάδα όσο το πολιτικό σύστημα δεν δέχεται να αντιμετωπίσει κατάματα την κατάσταση και το δημόσιο τομέα. Ζούμε μέσα σε μία περίοδο, αυτή την εποχή, μιας ψευδεπίγραφης Τη αισιοδοξία και εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται σιγά σιγά και καταγράφεται και στον τύπο και έξω από την Ελλάδα, ε, η οποία όμως δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αυτή η αισιοδοξία δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και αυτό το καλοκαίρι αναμένεται νέο κύμα φόρων που θα πλήξει την μεσαία τάξη, το καλοκαίρι επαναλαμβάνω, η, φορολογική, η βιομηχανική παραγωγή βρίσκεται σε πτώση παρά ε, την μικρή αυτή αύξηση των εξαγωγών. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει μια, έναν κικαιώνα ε, κακών δανείων, τοξικών δανείων. Οι εγγυήσει που έχουν δοθεί με τη μορφή των, έγκυων, των ε, εμπράγματων εγγυήσεων για να διασφαλιστούν τα δάνεια δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική ε, στήριξη και οι τράπεζες θα χρειαστούν περισσότερο κεφάλαιο. Περισσότερο κεφάλαιο λοιπόν για τις τράπεζες. Η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν εμφανίζεται στον ορίζοντα ακόμα και οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν με την ταχύτητα σαλίγκαρου. Κυρίε και κύριοι, η Τρόικα επέτυχε στην Ελλάδα την δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό το επέτυχαμε. Αυτό είναι μια επιτυχής προσπάθεια και κυρίως χάρη στον έλεγχο του, ε, της τσέπης του πολι... της Ελλάδας. Είτε θα κάνεις αυτό και θα ζώσουμε τα χρήματα, είτε αν δεν το κάνεις δεν θα έχεις χρήματα. Και έτσι αναγκάστηκε η Ελλάς να προχωρήσει τη δημοσιονομική προσαρμογή. Εκεί που απέτυχε όμως η Τρόικα ήταν να... στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα και αυτό για λόγους που ξεπέρνουν τη δική μου αντίληψη. Γιατί λοιπόν δεν τόλμησε να πιέσει πιο αποφασιστικά για μεταρρυθμίσεις. Την ευθύνη για τις μεταρρυθμίσεις την έχει αναλάβει η ομάδα δράσης, η Task Force. Δεν είχε όμως τα σχετικά μέσα επιβολής, τα μέσα επιβολής που είχε στη διάθεσή της από την άλλη πλευρά η Τρόικα για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Έτσι λοιπόν η Task Force εξαρτάται μόνο από την αναγνώριση και αποδοχή της κοινή λογικής για να γίνει, ε, για να φέρει πέρα στο έργο της. Δηλαδή, τη δύναμη της πυθούς. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό δεν φέρνει αποτελέσματα. Γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα σε σχέση με αυτήν την ιερή αγελάδα που βρίσκεται περιχαρακωμένη παντοχώθων. Η, ο, οι Έλληνε τώρα βρίσκονται χωρισμένοι σε δύο μεγάλε ομάδε. Αυτού που έχουν ε, χάσει ή που χάνουν τη δουλειά του και εκείνου που πληρώνουν φόρου. Μην ακούτε αυτά που σα λένε, τι ιστορίε, πληρώνουν φόρου οι Έλληνε και μάλιστα πολλοί πληρώνουν και πολύ υψηλού φόρου. Και υπάρχουν και αυτοί που μένουν στη δουλειά του, χάρη στα λεφτά που πληρώνει ο φορολογούμενος. Αυτή η κατάσταση όμω είναι αφόρητη, μακροπρόθεσμα είναι μη βιώσιμη και θα καταρρεύσει το σύστημα κάποια στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, μόνο 10 λεπτά ήταν η ομιλία μου. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε την ευκαιρία να δω, παρουσιάσω και ένα πρακτικό παράδειγμα που εμφανίστηκε χθε, που ταξίδευα για να έρθω στην Ελλάδα, ε, από την Ελλάδα εδώ. Πήρα λοιπόν την εφημερίδα Herald ε, Tribune. Στην πρώτη τη σελίδα είδα ένα άρθρο με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας το χάος του ελληνικού κτηματολογίου». Θα είδατε ίσως τις ε, καρτέλες της παρουσίασης του κυρίου Ράχενμπαχ, ίσως ήταν η δωδεκάτη καρτέλα από τις διαφάνειές του, ε, το, στο έργο που έχει να κάνει να επιτελέσει η ομάδα δράσης ήταν το κτηματολόγιο. Να σας πω λοιπόν το άρθρο γιατί ήταν πολύ ωραία η περιγραφή της ε, Herald Tribune. Να σας διαβάσω ένα κομμάτι. Και παραθέτω. Οι πιστωτέ, οι δανειστέ τη Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνέ Ορσματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχουν καταστήσει σαφές πως επιθυμούν την ανάπτυξη κτηματολογίου το ταχύτερο δυνατό. Και σχεδίου πόλεως το ταχύτερο δυνατό. Και συνεχίζω. Διεθνείς, διεθνούς προελεύσεως εμπειρογνώμενες έχουν επισκεφθεί το τελευταίο διάστημα την Ελλάδα, μάλλον αναφέρονται στην τάσκοση του κυρίου Ράχενβαχ, οι οποίοι κατέληξαν, έτσι λέει η Herald Tribune, ότι τα κύρια προβλήματα προέρχονται από ένα πολύ κακό σύστημα για την προμήθεια, ε, την ανάθεση που οδήγησε σε πολύ κακές ε, συμβάσεις. Μία δε από τις επιχειρήσεις, από τους εμπειρογνώμονες, ένας από τους εμπειρογνώμονες που έκανε αυτές τις διαρευνητικέ αποστολές από την Αυστρία, είπε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήθελε η κυβέρνηση να κάνει και πώς. Πολλά χρήματα δαπανήθηκαν χωρίς κανείς να γνωρίζει πού πήγαν τα χρήματα αυτά. Αυτά τα λέει ο κύριος Άρνηστα από την Αυστρία. Στόχος τώρα είναι να ολοκληρωθεί στο 2020. Άλλοι Έλληνες αξιωματούχοι αποκάλεσαν το στόχο αυτόν αισιόδοξο. Το 2013 μιλάμε και οι αξιωματούχοι Έλληνες λένε ότι το 2020 είναι υπεραισιόδοξο όταν περιμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Και για να ολοκληρωθεί θα έχει δαπανίσει 1,5 δις ευρώ η Ελλάδα προκειμένου να τακτοποιήσει την κατάσταση. Να συγυρίσει τα πράγματα. Αυτό είναι το χθεσινό άρθρο της Herald Tribune. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλά χρήματα, δικά σας χρήματα, έχουν δαπανηθεί. Κανείς δεν γνωρίζει που πήγαν. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα 100% χαρακτηριστικό. Αυτό το κτηματολόγιο, ένα μεγάλο έργο, να κάνουμε ένα μεγάλο έργο, να κάνουμε το μεγάλο αυτό κτηματολόγιο, πολύ ωραία, ναι βεβαίως να το κάνουμε, το αναθέτουμε όμως σε ένα δημόσιο τομέα της Ελλάδας, ο οποίος είναι σε απόλυτη ανικανότητα να το επιτελέσει, να το εκτελέσει και είναι και σε απόλυτη άρνηση να το εκτελέσει. Δεν θέλει, δεν έχει ενδιαφέρον να το εκτελέσει. Δεν θα εξηγήσω γιατί δεν θέλουν το κτηματολόγιο κάποιοι, αλλά είναι αλήθεια ότι δεν το θέλουν. Χάνονται πολλά χρήματα, δικά σας χρήματα. Κάποιοι γίνονται πλούσιοι, άλλα ερωτηματικά εκεί, και εν τέλει τίποτα δεν γίνεται. Και το πρόβλημα με το κτηματολόγιο στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ σοβαρέ συνέπειες. Πάρα πολύ σοβαρές. Πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει τι είδου φόρο θα επιβάλλει στην ε, περιουσία, όταν δεν γνωρίζουμε ποιο έχει τι στην κυριότητά του. Επιπλέον, το γεγονό αυτό και παρόλα αυτά δεν έχει εμποδίσει την Τρόικα, η οποία ανοήτως πως επιμένει να επιβληθούν φόροι εκεί που δεν υπάρχει το θεματολόγιο. Όταν μας λέει η Τρόικα, η Τρόικα επιβάλλεται φορό περιουσίας, μα δεν έχουμε βάση πάνω στην οποία να μπορέσουμε τεχνικά, πρακτικά να επιβάλλουμε το φόρο. Μερικές φορές δίνεται η εντύπωση λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι της Τρόικα είναι απλώς ε, χαρτογιακάδες οι οποίοι μετράνε νούμερα, τα γράφουν, τα βγάζουν και πιστεύουν ότι με το να γράψουν τα νούμερα κάτι θα γίνει. Ε, όχι, δεν γίνεται λοιπόν. Ένα πρακτικό λοιπόν συμπέρασμα, μια πρακτική λύση και το, την απευθύνω στον κύριο Ράχενμπαχ θα ήταν η εξή. Κόφτε το πρόβλημα σε πιο πολλές μικρές φέτες. Ξεκινήστε με προτεραιότητα, προτεραιότητες. Πείτε πρώτα αστικά κέντρα, μεγάλα αστικά κέντρα. Μην πιάσετε να κάνετε όλη την Ελλάδα. Πιάστε τα, ε, σε μικρότερες φέτες τα αστικά κέντρα που είναι το το 5% ίσως του συνόλου, αλλά ίσως να προσωπούν το 90% της συνολικής αξίας της γης. Ξεκινήστε λοιπόν με ένα μικρό κομμάτι, αλλά υλοποιήστε το αυτό το μικρό κομμάτι, ολοκληρώστε το. Και έκανα πρόσφατα μια πρόταση εγώ ίδιο στην κυβέρνηση, αλλά δεν με ακούνε. Ένα εκατομμύριο ευρώ και έξι μήνες μόνο θα αρκούσαν για να καταγράψουμε την επιφάνεια οικοδομημένων οικοπαίδων σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας και με βάση αυτή τα, αυτά τα στοιχεία μπορούμε να φτιάξουμε ένα απλό, σαφές, αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα με βάση το οποίο ο καθένας θα πληρώνει τους φόρους του. Δυστυχώ όμω αρχίζουμε με μεγάλα σχέδια, χανόμαστε μέσα σε αυτά, χάνουμε τα λεφτά μα και τελικά δεν γίνεται τίποτα. Επιπλέον θα μπορούσαμε με αυτό το κτηματολόγιο στο οποίο αναφέρομαι να περιορίσουμε το πρόβλημα ακόμη περισσότερο. Εάν εστιαζόμασταν σε ένα μεγάλο Δήμο. Θεσσαλονίκη, Φερρυπίν ένας ε, Δήμος που έχει ένα πολύ προοδευτικό δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε αυτό το Δήμο για να προχωρήσουμε το έργο του κτηματολογίου. Και γι' αυτό απευθύνομαι πάλι στον κύριο Ράχινμπαχ λέγοντα, ε, αντί να πιάνουμε τα μεγάλα έργα και τι μεγάλε προθέσει, α κάνουμε πιο, μικρές, ε, πιο μικρά σχέδια, πιο περιορισμένου ελληνικού, αλλά α τα ολοκληρώσουμε γιατί οτιδήποτε τελειώσει γίνεται και ένα καλό παράδειγμα προ και επίσης μην δίνετε συμβουλές, πράξετε, πράτετε. Θα θυμίσω μια ιστορία, κάποιος που θέλει να μάθει να, να παίζει ε, μπάσκετμπολ, καλά, ρώτησε μα πώς θα μάθω. Ε, του λένε κοίτα πώς παίζει ο Τζόρνταν. Μα δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε από κάποιον να κάνει κάτι όταν δεν είναι σε θέση να το κάνει πρέπει μόνος του να βρει τον τρόπο να το, κάνω, να το κάνει. Αυτή θα ήταν η συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω εάν ζητούσε κανείς τη συμβουλή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μάνο. Στην πραγματικότητα 21 λεπτά μιλήσατε, αλλά βέβαια ήταν πολύ σημαντικό ε, και έχουν ζητήσει διάφοροι το λόγο για να ε, σχολιάσουν να δώσουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις παρουσιάσεις και να περάσουμε λοιπόν στη συνέχεια στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον ε, κύριο Νόρμουντ Σποέν, ε, ε, αναπληρωτή Γενική Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζο. Έχετε το λόγο και έχετε 15 λεπτά για να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Δικό μου καθήκον σήμερα είναι να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή του Ταμείου Συνοχής ε, και των σχετικών κονδύλιων στην Ελλάδα. Θα επικεντρωθώ λίγο στο ε, στην κατάσταση σήμερα, το τι ακριβώς κάναμε εμείς για να ανταποκριθούμε στην κρίση από πλευράς πολιτικής, τις βασικές προκλήσεις και επίσης θα επικεντρωθώ λίγο και στο μέλλον ε, στην παρουσίασή μου, διότι όπως είπαμε σήμερα υπάρχει πλέον ένα παράθυρο ευκαιρίας, ε, διότι προγραμματίζουμε την επόμενη επταετία από το 2014 και τούδε και νομίζω ότι υπάρχουν κάποια διδάγματα τα οποία έχουμε αντιλήσει και έχουν γίνει και πάρα πολύ ε, σημαντικά πράγματα και το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Ε, να πω λοιπόν καταρχάς ότι για την Ελλάδα ε, προβλέπονται άνω των 20 δισεκατομμυρίων από πλευράς πολιτικών συνεχής από το 2011 μέχρι το 2013 και στόχος είναι να βοηθήσουμε τον εξυγχρονισμό των υποδομών της χώρας, να μειώσουμε την ανισότητα των περιφερειών και να προωθήσουμε την εδαφική συνοχή και την κοινωνική συνοχή. Ε, μέχρι τούδε άνω του 56% των κονδυλίων ε, από το Ταμείο Συνοχής έχουν ε, διατεθεί ε, κυρίως από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής που είναι τα ταμεία τα οποία διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο και αυτό το ποσοστό του 56% είναι λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δείτε όμως τι επενδύσεις έχουμε κάνει, είναι όλες πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία. Έχουμε χρηματοδοτήσει προγράμματα μεγάλης κλίμακας, αλλά μέχρι και προγράμματα χαμηλότερης ε, τοπικής κλίμακας. Όλα όμως είναι εξίσου σημαντικά για την αναβίωση της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επομένως εδώ έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν εγκριθεί για προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και έχουμε ε, ήδη εκταμιεύσει 55% αυτών των κονδυλίων και επομένως πάνω από 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούμε ότι έχουμε υποφοληθεί από αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν επίσης και κάποιες επιτυχημένες ε, περιπτώσεις στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη η κοράλια στον τομέα των μικροελεκτρονικών ε, και μπορούμε να αναφέρουμε αυτές τις επιτυχημένες περιπτώσεις και θα πρέπει να το κάνουμε διότι δεν έχουμε μόνο άσχημες ιστορίες για την Ελλάδα. Το βασικό για μας βέβαια είναι και επενδύσει σε υποδομές, σε δίκτυα κυρίως, ε, να άρουμε τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις μεταφορές. Επίσης ε, να πω ότι μας ενδιαφέρουν αυτά ε, τα προγράμματα υποδομών γιατί ε, σε αυτά έχουμε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ η επέκταση του μετρό της Αθήνας η ανάπτυξη του μετρό της Θεσσαλονίκης και κάποια θέματα τα οποία ανέφερε σήμερα ο κύριος Ράιχινμπαχ για τις οδικές υποδομές και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα και να ολοκληρωθούν εκτίμηση είναι ότι από τα ταμεία δημιουργούνται πάνω από 140.000 θέσει εργασία στην Ελλάδα και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τι γίνεται με τις ε, διαρθρωτικές ε, επενδύσεις. Θεωρώ ότι τα διαρθρωτικά κονδύλια είναι ίσως τα βασικά εργαλεία για να δώσουμε νέα όθηση στην ε, ανάπτυξη και φυσικά στην απασχόληση στην Ελλάδα. Τα ταμεία λοιπόν είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικά στην Ελλάδα και αυτές είναι πραγματικές επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση. Αν δείτε τι ακριβώς έχουμε επιτύχει, διότι όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα ήταν σαφές ότι χρειάστηκε να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή σε κάποια θέματα και να σχεδιάσουμε και κάποια νέα στοιχεία για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ε, ε, τις πολιτικές μας και να επενδύσουμε τα κονδύλια μας. Ε, ήδη ευθύ εξ αρχής είχαμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια προσκόμματα στην Ελλάδα σε θέματα εφαρμογής, αλλά βοηθήσαμε τη συνεργασία, την εντατικοποιήσαμε και φυσικά ε, ε υιοθετήσαμε και μία πιο απτή προσέγγιση και να υπάρχει πιο στενή παρακολούθηση και συνεργασία με την ε, ε, ελληνική κυβέρνηση και φυσικά με την σύσταση της Task Force είδαμε ότι έγιναν κάποια σημαντικά βιάματα για την άρση των προσκομμάτων. Ε, κάποια παράδειγματα, ο Επίτροπος Χάν το 2011 ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να καθορίσει έναν κατάλογο 181 προγραμμάτων προτεραιότητας όπως για παράδειγμα τις συμβάσεις παραχώρησης. Κάποια εξ αυτών τα ανέφερε ο κ. Ράχεν Μπαχίδη και αυτά είναι προγράμματα τα οποία είναι υψής της σημασίας για την ανάπτυξη ανάπτυξη της ε, Ελλάδος ε, θα βοηθήσουν την ελληνική ε, οικονομία και θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. Γι' αυτό ακριβώ και παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων. Ε, με τα χαράς διαπιστώνουμε ότι έχει φτάσει και κατάλληλη στιγμή για τις συμβάσεις παραχώρησης για τα οδικά δίκτυα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η χρηματοδότηση είναι άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και σίγουρα θα δημιουργηθεί ουσιαστικός αριθμός ευκαιριών απασχόλησης. Γι' αυτό ακριβώς είναι και πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα προγράμματα να εφαρμοστούν καταλήλως. Ε, δεύτερον, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, καταπολέμηση της ανεργίας, ε, ιδίως ε, διότι ο πρόεδρος Μπαρόζο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ε, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για τους νέους το 2012 και επομένω ε, σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα αναπτύξαμε ένα σχέδιο δράσης για να δώσουμε όθηση στην επιχειρηματικότητα και να αυξήσουμε την απασχόληση για τους νέους. Και εδώ έχουμε λοιπόν άνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει όμως ένα πρόγραμμα δράσης και αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε τώρα είναι ότι θα εφαρμοστεί. Ε, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των ε, διαρθρωτικών ταμείων ε, και τις επενδύσεις για το μέλλον και την Ελλάδα και στην Ελλάδα υπάρχει και ένα μνημόνιο συνεννόησης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Εντό αυτού του μνημονίου συνεννόηση αντανακλάται όλη η πολιτική συνοχή. Υπάρχουν συγκεκριμένα ορόσημα τα οποία σχετίζονται με την πολιτική συνοχή, καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι ανά ε, μας ενδιαφέρει αναθεώρηση τη νομοθεσία για τι κρατικέ προμήθειε, ολοκλήρωση των προγραμμάτων, να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή ε, στρατηγικής καταπολέμησης της απάτης και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την πολιτική συνοχή και περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Ε, επίσης θα ήθελα να ε, σταθώ και στην απλούστευση της νομοθεσίας και των διαδικασιών. Ε, εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και ο Επίτροπος ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να αναθεωρήσουν την κατάσταση, γιατί αν δείτε πώς έχει κατάσταση στα κράτη-μέλη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιπλοκές σε επίπεδο κρατών μελών για τις πληρωμές, τους δικαιούχους, την επιλογή των προγραμμάτων, αλλά επίσης και πολλές άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εδώ θα πρέπει να πω ότι η ελληνική Task Force έχει βοηθήσει ιδιαίτερα και έχουν ε, δώσει όθηση στους τομείς αυτούς ε, και η επίτευξη των στόχων αυτών βεβαίως περιλαμβάνεται και αυτή στο Μνημόνιο Συνεννόησης. Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη ε, προσοχή σε τομείς τους οποίους καθυστερούμε, όπως για παράδειγμα στην ε, περίπτωση του περιβάλλοντος, ε, στη διαχείριση των αποβλήτων. Εδώ συνεργαζόμαστε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με τις ελληνικές αρχές για να ε, διαχειριστούμε το πρόβλημα. Έχουμε επίσης κάνει μια αναδιάταξη στο πρόγραμμα, έχουμε δει τι απομένει και έχουμε ένα ποσό ενός δισεκατομμυρίου το οποίο θα διατεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα μέσα ε, χρηματοοικονομική στήριξη, διότι όταν δεν χρηματοδοτεί κατάλληλα ο τραπεζικός τομέας, ε, δημιουργούνται προβλήματα για πάρα πολλού οικονομικούς φορείς. Γι' αυτό ακριβώ λοιπόν δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή για την ενίσχυση της χρήση των κατάλληλων μέσων ε, στην Ελλάδα. Έχουμε προτείνει και στη συνέχεια ενεκρίθησαν και συγκεκριμένες διατάξεις για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ε, ε, δυνατότητες. Ε, κάποια ταμεία όπως το Jeremy για παράδειγμα λειτουργούν αποτελεσματικά, έχουν διατεθεί κονδύλια σε μικρές επιχειρήσεις ως κεφάλαιο κίνησης και επίσης όπως ανέφερε και ο Χόρς Ράιχενμπαρχ, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία, να ε, ε, διαθετεθεί αυτό το 1 δισεκατομμύριο για τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις ε, και πρέπει να φροντίσουμε να ξεκινήσει η διάθεση των κονδυλίων το συντομότερο δυνατόν. Να σας πω δε ότι αυτή είναι η αρχή και μόνον αυτής της εκλογήκευσης των μέσων. Στόχος είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος όπου το ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτά τα μέσα θα είναι πιο ισχυρό, πολύ πιο ενδελεχές και πολύ πιο αποτελεσματικό. Τέλος, πρέπει να σας πω ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι μεν 56% αλλά ταυτόχρονα έγινε και προσαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης λόγω της κρίσεως και ε, ε το κατανοούμε αυτό. Κάναμε μια πρόταση και έγινε αποδεκτή για την Ελλάδα. Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης είναι 85% και υπάρχει και ένα πρόσθετο 10% για την περίοδο της χρηματοοικονομικής βοήθειας. Ε, ξέρω ότι περνάει ο χρόνος, αλλά θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τις βασικές προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον. Το 2013 είναι κρίσιμο έτος, διότι πρέπει να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι το 2015 για να ολοκληρωθούν ε, κάποια προγράμματα. Αλλά η ολοκλήρωση προγραμμάτων που εκκρεμούν είναι ακόμα μεγάλη πρόκληση. Προσπαθούμε λοιπόν εντός του 2013 να περατωθούν κάποιες συμβάσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής ή να είναι ήδη ανεξελίξη. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά και πρέπει να επικεντρωθούμε και στην εφαρμογή και στις πληρωμές. Γι' αυτό και έχουμε θέσει στους στόχους για το Μνημόνιο Συνεννόησης ε, υπάρχει ένα ποσό 3,890 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρέπει να δαπανηθεί από τα ταμεία συνοχής, που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και πάρα πολύ στενή παρακολούθηση της εφαρμογής. Η Ελλάδα θα χρειαστεί λοιπόν σε 2,5 χρόνια να δημιουργήσει αυτό το 50% των δαπανών που ε, ε μας απασχολούσαν τα τελευταία χρόνια. Η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να πω και δύο λόγια για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι εν εξελίξη, υπάρχουν διστάμενες απόψεις για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά κατά την άποψή μας ε, για όλους όσους ασχολούνται με την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων, είναι σαφές ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει κατεπηγόντως να αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Ε, καθυστερήσεις που αφορούν την οριμότητα των προγραμμάτων, καθυστερήσεις αδειοδοτήσεις, έλλειψη ρευστότητας και έλλειψη αφήνεια σε κάποιες διαδικασίες είναι από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να επιλύσουμε γρήγορα. Όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης και της ιδιοκτησίας από τις ελληνικές αρχές, εξακολουθεί να εκκρεμεί το θέμα του συντονισμού ε, μεταξύ Υπουργείων και κάποιων περιφερειακών αρχών και αυτό είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις. Και τέλος φυσικά πρέπει να υπάρχει η η καταπολέμηση της διαφθοράς με μέτρα καταπολέμησης τη διαφοράς είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εφαρμογή των ταμείων και φυσικά θα δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Ο Επίτροπός μας θα πάει και στην Ελλάδα τον Οκτώβριο για να μιλήσει για την καταπολέμηση της απάτης και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να πω ότι δεν υπήρξαν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα ποιότητα των δαπανών, γιατί οι δομέ είναι αρκετά ισχυρέ, έχουμε μακρά πείρα. Υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά στι κρατικέ ενισχύσει, παραδείγματι, αλλά δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα προ το παρόν. Τώρα για το μέλλον, γιατί ξεκινάει ο σχεδιασμός ε, για τα προγράμματα από το 2014 στο 2020. Είναι μια νέα δομή και όπως έχουμε πει σε όλα τα κράτη-μέλη παντού και πάντα, δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα κάνουμε ως συνήθως. Έχουμε αντλήσει τα διδάγματά μας, γνωρίζουμε τι είναι καλύτερο, σας τα έχουμε αναφέρει και εσάς ε, αρκετές φορές, ε, πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις στην εφαρμογή των ταμείων. Και είναι σαφές ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά ε, και πιο επικεντρωμένα σε αποτελέσματα όλα όσα κάνουμε και γι' αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη στον άτυπο διάλογο για το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων υποδομών και να έχουμε επενδύσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, η ευφυής εκδίκευση και τέλος να δώσουμε μια όθηση στην απασχόληση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε και η Ελλάδα Ελλάδα να επικεντρωθεί σε ένα περιορισμένο αριθμό ενωτήτων θεματικών που ε, επιτρέπονται μέσω της νομοθεσίας και πρέπει φυσικά να επιλέξουμε τι θα χρηματοδοτούμε και τι δεν θα χρηματοδοτούμε στο μέλλον. Χρειαζόμαστε την κρίσιμα μέσα βέβαια των επενδύσεων και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Και θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε και κάποιες ε, αβάσταχτες οικονομικές δομές στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα πάσχει σε κάποια θέματα ε, όπως ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, ε, κατάλληλες προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις, διοικητικές και νομικές διαδικασίες που είναι πάρα πολύ περίπλοκες και αυτά φυσικά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφύσισε να αναλάβει πιο δραστηριό ρόλο στο μέλλον. Συνεργαστήκαμε και με άλλες υπηρεσίες Έχουμε ετοιμάσει και τα έγγραφα για την κάθε χώρα και εδώ έχουμε εντοπίσει και τις βασικές προκλήσεις στα κράτη-μέλη και αντιστοίχως έχουμε προτείνει και κάποιες προτεραιότητες χρηματοδότησης για κάθε κράτος μέλος. Για την Ελλάδα η πρώτη πρόκληση είναι το οικονομικό μοντέλο το οποίο δεν είναι πλέον βιώσιμο διότι δεν έχει ανταγωνιστικότητα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να υποστηρίξουμε τις καινοτομίες, ένα φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Η ανεπαρκής δημόσια διοίκηση είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ευνοήσουμε για τη χώρα. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε λοιπόν και να αναβαθμίσουμε την εικόνα της δημόσιας διοίκηση, δηλαδή να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες, υπηρεσίες προς τους πολίτε και τις επιχειρήσεις. Μας ενδιαφέρει επίση το θέμα των υποδομών. Πρέπει να συνεχίσει ο εξυγχρονισμό των υποδομών, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα στρατηγικό πλαίσιο οικονομική ανάπτυξη τη χώρα και όχι ε, με μονομένη χρηματοδότηση ε, προγραμμάτων που δεν έχουν καμία συνέπεια. Τέταρτον, ανεπαρκή χρήση φυσικών πόρων και αλλαγή του κλίματο, δηλαδή θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. ε, ε, ασφάλεια εφοδιασμού και τέλος κάτι εξίσου σημαντικό η υψηλή ανεργία και η αυξηνόμενη ε, ένδια και κοινωνικός αποκλισμός και φυσικά ο συνάδελφος ε, θα πει για κάποια πράγματα γι' αυτό εντός ολίγου. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου θα ήθελα να σας πω ότι εξετάσαμε πάρα πολύ σοβαρά ε, κάποιες λύσεις για το μέλλον προς την επιτυχία για το επόμενο διάστημα, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, κατάλληλη ε, συγκέντρωση, το να επικεντρωθούμε σε ποιοτικέ δαπάνες, ε, να αναλαμβάνονται ταυτόχρονα οι κατάλληλε ευθύνε, όλα αυτά αποτελούν ε, κλειδί για την επιτυχία. Και φυσικά όπω γνωρίζετε προκειμένου ότι επιτύχουμε αυτό και είμαστε ευγνώμονε προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το υποστηρίζει και το Συμβούλιο, την εκ των προτέρων ερωσιμότητα. Δηλαδή δεν θα χρηματοδοτήσουμε καμία προτεραιότητα επενδύσεων εάν δεν πληρούνται οι κατάλληλε προποθέσει. Και αυτό για την Ελλάδα ε, σημαίνει και θα ήθελα να το αναφέρω ε, η στρατηγική για παράδειγμα της εφιούς εξειδίκευσης ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει κατάλληλο πεδίο για καινοτομίες και αυτό θα είναι λοιπόν μια ε, από τις προϋποθέσεις που θα θέτουμε εκ των προτέρων. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, φιλικότερες δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επίσης μεταφορά ε, της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κυρίως για την διαχείριση των αποβλήτων και ούτω καθεξής ε, πρέπει να σας πω ότι θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα παρακολουθήσουμε στενά την εφαρμογή αυτών των όρων που θα τίθενται εκ των προτέρων και να σας πω ότι το, ε, η μη εφαρμογή θα σημαίνει ότι θα αναστέλλονται και οι πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή έχει μακρά πείρα στην εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και όπως σας είπα οι δομές εφαρμογής είναι πολύ ισχυρές και υπάρχουν άτομα με κατάλληλες δεξιότητες και αυτό λοιπόν θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει αυτό και θα βασιστούμε και στα διδάγματα που αντλήσαμε στο διάστημα αυτό. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προοδεύει. Ε, βλέπουμε ότι βελτιώνονται σταθερά τα οικονομικά, ο ε, πεζικός τομέας προχωρά με την ανακεφαλαιοποίηση και ε, φυσικά προχωρούν και κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερο από ποτέ πρέπει πλέον η πολιτική συνοχή να επικεντρωθεί σε μέτρα ανάπτυξης και να υποστηρίξει πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στην Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις μας στην ανάπτυξη καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνουμε και τη σημασία της παιδείας, και των ε, συστημάτων ε, ε, κατάρτισης, δηλαδή όλα αυτά θα είναι αλληλένδετα και θα διέπουν τις οικονομικές δραστηριότητες. Και όλα αυτά φυσικά ε, σημαίνει ότι θα έχουμε και κατάλληλες επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Και εμείς από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης ε, Ρέτζο ε, και η Task Force, ε, όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης θα βοηθήσουμε την Ελλάδα για να μπορέσουμε να αναβιώσουμε την ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. 19 Σας ευχαριστώ πολύ. 19 <clears throat> λεπτά κράτηση ομιλία σας. Παρακαλώ τον επόμενο μιλητή να περιοριστεί στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε ορίσει, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ε, δώσουμε χρόνο για συζήτηση. Ο κύριος Στάπ Γιώργενσεν από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζει η παρουσίαση δηλαδή. Παρακαλώ. Please. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε δυνατόν πιο σύντομο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε έδωσα μόνο μία διαφάνεια για την παρουσίασή μου. Η διαφάνεια που βλέπετε εκεί πάνω στην οθόνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το μέσον για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Είναι το εργαλείο που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας, το συγκεκριμένο δηλαδή μέσο, είναι να επενδύουμε στον άνθρωπο με τέσσερα λειτουργικά προγράμματα. Βλέπετε συγκεκριμένα στην οθόνη το μεγαλύτερο, το πρώτο, η μεγαλύτερη στήλη, το λειτουργικό πρόγραμμα για τους ανθρώπινους πόρου. 2,8 δις ευρώ έχουν δαπανηθεί για την προσαρμογή των δεξιοτήτων, προσόντων, ικανοτήτων των ανθρώπων ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται σε μια πιο παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά. Και αυτό το πράττουμε ιδιαίτερα με μέρημνα για τις πιο ευάλωτες ομάδες της αγοράς εργασίας, εκείνες που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας περίπου, και εκείνες που χρειάζονται να βρουν και να διατηρήσουν μια θέση εργασία. Επενδύσεις επίση έχουμε στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα τη ψυχικής υγεία που καλύπτει το πρόγραμμά μας. Ένας από τους προλαλήσαντε είπε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα στις περιφέρειες. Δεν φτάνουν στον άνθρωπο. Τα λειτουργικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου νομίζω ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι έχουν αγγίξει τις ζωές 3 έως 3,5 εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτή την περίοδο. Είμαστε γνωστοί, έχουμε μεγάλη αποδοχή στα έργα μας και στα προγράμματά μας. Το δεύτερο λειτουργικό πρόγραμμα που βλέπετε στη δεύτερη στήλη είναι το λειτουργικό πρόγραμμα για την ε, παιδεία και την διαβίου μάθηση. 1,7 δις ευρώ θα πανώνται για το λειτουργικό αυτό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας, την κοινωνική ε, συμπερίληψη ενσωμάτωση ώστε να μπορεί κανείς να μπαίνει στην αγορά εργασίας με την διαβίου μάθηση η οποία σημαίνει να βελτιώνει κανείς διαρκώς και να διατηρεί τις δεξιότητες και τις γνώσεις του και εκείνη η προτεραιότητά μας με την, ε, ε, με κύριους άξονες και την επαγγελματική κατάρτιση αλλά και τη δυνατότητα να βρει κανείς το δρόμο για να μπει στην αγορά εργασίας. Στο τρίτο πρόγραμμα, τρίτη στήλη της διαφάνειας, βλέπετε το λεγόμενο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης. Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ανοίγματο πνεύματος, της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Και αυτό το λέω σε επίπεδο κεντρικής, κεντρικό, κεντρικής κυβέρνησης γιατί το πρόγραμμα καλή κράτης δεν το καλύπτουμε εμείς. Ε, ήταν δύσκολη η εφαρμογή αυτού του προγράμματος, του λειτουργικού για την κεντρική διοίκηση. Αντιμετωπίσαμε εμπόδια κυρίως τα χρόνια της κρίσης είναι δύσκολο βεβαίως να γίνει μεταρρύθμιση και των διοικητικών δομών. Πρόκειται λοιπόν για αυτό το ε, λόγο για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη αναδιατυπωθεί, αναδιαμορφωθεί για να προσαρμοστεί στην κρίση. Προχωρεί τώρα. Η πορεία του είναι ήδη καλή και ελπίζουμε ότι θα δώσει αποτελέσματα σε αυτή την προγραμματική περίοδο για την οποία έχει προβλεφθεί. Το τελευταίο δε πρόγραμμα είναι ειδικού χαρακτήρα, πρόκειται για ένα ειδικό αποθεματικό ανάγκης, δηλαδή για μια περίοδο δύσκολη, στην αρχή της προγραμματικής περίοδου, βάζουμε στην άκρη χρήματα για να τα αξιοποιήσουμε όταν χρειαστεί. Η δύσκολη περίοδο βέβαια στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι ήδη είναι εν εξελίξη. Αξιοποιούμε λοιπόν τα κονδύλια αυτά για να στηρίξουμε όπου χρειάζεται 250 εκατομμύρια ευρώ για την επιχειρηματικότητα, για την επαγγελματική καθοδήγηση σε ανέργους, για το, ε, από τον χώρο της Λιανικής, από το χώρο των αντιπροσωπιών αυτοκινήτων και από άλλους τομείς που χρειάζονται επαναπροσανατολισμό. Για δε την Επιτροπή σας, ιδιαίτερα πιστεύω, ενδιαφέρον, θα έχει το επίπεδο της, ε, ε της ανάθεσης των δεσμεύσεων δηλαδή που έχουμε επιτύχει. Για τα λειτουργικά μας προγράμματα έχουμε επιτυχία 86% στις αναθέσεις για το πρώτο, για τους ανθρώπινους πόρους, 93% για την παιδεία και λίγο χαμηλότερα ποσοστά για τα δύο μικρότερα προγράμματα. Αυτά, αυτή η εικόνα λοιπόν αντικατοπτρίζει δύο στοιχεία. Καταρχάς ότι έχουμε προσαρμόσει τα προγράμματα στην κατάσταση της κρίσης. Προχωρούν συντονισμένα, ε, συγχρονισμένα με την κρίση τα προγράμματα αυτά και βοηθούν την ελληνική κυβέρνηση να, ε, να ανοίξει το δρόμο για τη διέξοδο από την κρίση. Ήδη πέρσι κάναμε μια μεγάλη αναδιατύπωση των προγραμμάτων αυτών και των τεσσάρων μεγάλων προγραμμάτων για να ενσωματώσουμε και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων σε αυτά. Προσαρμόζουμε δηλαδή τα λειτουργικά μας προγράμματα στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε μέσα στη χώρα. Και επιπλέον, από το ρυθμό αυτής της υλοποίησης θα δείτε ότι η Ελλάδα έχει καλά αποτελέσματα, πολύ καλά αποτελέσματα στην απορρόφηση κονδυλίων στους δύο κύριους τομείς που έχουμε εντοπίσει. Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση Ελλάδος έχει αντίληψη πλήρη των προκλήσεων που έχει στο μέλλον να αντιμετωπίσει. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την ε, ομάδα ε, δράσης, είμαστε σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση και για τα περιφερειακά και είμαστε σε θέση να διαφυλάσσουμε την σωστή εφαρμογή των διευθυντικών ταμείων και των κονδυλίων τους και σταματάω εδώ χωρίς να έχω ξεκλείσει ούτε 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την πάρα πολύ πλήρη παρουσίασή σας. Ο κ. Πλέκναπεν είναι ο επόμενος ομιλητής της Ευρω... Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να εξηγήσω λίγο τι κάνει η τράπεζά μας ε, στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες και την συρρήκνωση, την ύφεση στην ελληνική οικονομία τα τελευταία πέντε χρόνια, 6% περίπου το χρόνο, 25% για αυτήν την πενταετία. Η κατάσταση λοιπόν είναι δύσκολη και δύσκολο είναι και να βρει κανείς καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και φυσικά έχει πληγεί η αξιοπιστία, η χρηματοληπτική και την ίδια ώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν νέες πηγές χρηματοδότησης. Μειώνεται σημαντικά το επίπεδο επενδύσεων στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν έχουμε συμπεριλάβει στις ε, προσπάθειές μας στην εξέβρεση αυτής της χρηματοδότησης και βεβαίως τεχνική βοήθεια. Προσπαθούμε να βρούμε νέα μοντέλα, νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι σήμερα πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει πολλά και είμαστε κοντά στην ε, εξέβρεση πραγματικής χρηματοδότησης ε, για προγράμματα τα οποία ξεκινήσαμε. Υπάρχει ένα ταμείο εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις πολύ σύντομα, πιστεύουμε. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στην χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Μπορούμε να συνεισφέρουμε μέχρι και με ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Ήδη 225 εκατομμύρια ευρώ έχουν ε, ενσωματωθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των ελληνικών τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προτείνει ένα ε, σχέδιο το οποίο θα υπογραφεί στις 12 Ιουνίου για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης του εμπορικού τομέα. Πρόκειται για το Trade Finance Scheme. Όπως ξέρετε, οι ελληνικές τράπεζες χρηματοδοτούν και εμείς είμαστε ο εγγυητής. 500 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σχήμα και το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και 1-1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου, εμείς προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην χρηματοδότηση των παραχωρήσεων μεγάλων προγραμμάτων συνοχής, όπως παραδείγματος χάρη ε, η αυτοκινητόδρομη, ουσιαστικό πρόγραμμα Έχουμε ήδη συνεισφέρει με 650 εκατομμύρια ευρώ. Βρισκόμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Οι συμβάσεις θα υπογραφούν, πιστεύουμε, πριν την αρχή του καλοκαιριού. Και βεβαίως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 20.000 νέες θέσεις απασχόλησης άμεσα ή έμεσα και περίπου 0,3% αύξηση του ΑΕΠ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, αν τις ε, προσθέσουμε, βλέπετε ότι το Ταμείο Εγγύσεων, αυτό το σχήμα για την χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών, καταλήγουν σε ένα σύνολο επενδύσεων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που έχει σαν σκοπό να αντιστρέψει την τάση της ύφεση. Επίσης έχουμε δεσμευθεί για άμεσες χρηματοδοτήσεις για 200 εκατομμύρια ευρώ για τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Πάτρα που πιστεύω ότι πολύ σημαντικές επιπτώσεις, θετικές επιπτώσεις θα έχει στην πραγματική οικονομία. Μέχρι το μέσο του 2013 θα έχουν εκταμιευθεί περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Στοχεύουμε μετά από τις υπογραφές που θα οδηγήσουν σε εκταμιεύσεις, γιατί η υπογραφή είναι το πρώτο στάδιο πριν την ε, εκταμίευση. Στοχεύουμε λοιπόν να φτάσουμε το 1 ή 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 2013. Ήδη το διοικητικό μας ε, συμβούλιο έχει εγκρίνει 400 εκατομμύρια για το μετρό της Θεσσαλονίκης και συμβάσεις παραχώρησης για άλλα προγράμματα τα οποία έχουν προχωρήσει σημαντικά και θα ευοδοθούν κατά την άποψή μας πολύ σύντομα. Ο εισηγητής, ο κύριος Χατζημαρκάκης, εξέφρασε κάποιες ανησυχίες. Συμφωνούμε με τις ανησυχίες που εκφράσατε. Συμφωνούμε ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν, ότι συνεχίζει να υπάρχει δυσπραγία και αδυναμίες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Εμείς σαν τράπεζα ανασχεδιάσαμε τον τρόπο παρέμβασής μας, το πρότυπο παρέμβασής μας, με σκοπό να δραστηριοποιήσουμε την παρέμβασή μας όχι απλώς χρηματοδοτώντας, αλλά στηρίζοντας. Επαναλαμβάνω ότι επιθυμούμε με την τεχνική βοήθεια που παρέχουμε στην Ελλάδα να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βελτιώσει τη διαρθρωτική της δυσκολία υπάρχουν θέματα διακυβέρνηση, παραδείγματο χάρη. Προσπαθούμε λοιπόν και σε αυτά να ε, συνεισφέρουμε στη βελτίωσή τους. Σαν τράπεζα, λοιπόν, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας, γιατί όπως ξέρετε, το τριπλό α, το οποίο έχουμε σήμερα σαν τράπεζα από τους οίκους αξιολόγησης, εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας κάθε φορά που παρεμβαίνουμε ε, σε μια χώρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ που κρατήσατε και το χρόνο σας. Και μια και έχουμε το χρόνο, μπορούμε τώρα να ακούσουμε τους επτά συναδέλφους που έχουν στήσει το λόγο Έχουμε 47 στη θέση μας, 47 λεπτά στη θέση μας. Αν θέλετε... και ο κύριος Αντί. Λοιπόν, 5 λεπτά το πολύ ο καθένας παρακαλώ. Και καλό πρώτον, πρώτην, την κυρία Αγιάλα Σέντερ να λάβει το λόγο, αν και τη βλέπω να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορείς τώρα, Ινές? Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν ήξερα ότι ήμουν πρώτη-πρώτη στον κατάλογο των ομιλητών. Ήθελα απλώς ε, προς το παρόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Ράχενμπαχ. Ε, ε, λυπάμαι βέβαια που δεν είναι εδώ. Ίσως θα... να είναι κάποιος εδώ ο οποίος θα σημειώσει τις ερωτήσεις για να του ε, τις θέσουμε. Θα ήθελα Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη, σας έψαχνα πιο μπροστά, εκεί συνήθως έχουμε τις εκπροσώπους της Επιτροπής και δεν σας είδα. Ε, χαίρομαι που είστε ακόμα εδώ. Ήθελα, επειδή προέρχομαι και από μια χώρα την Ισπανία, η οποία και αυτή ε, έχει μπλεχτεί στα γενικότερα προβλήματα και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το τι συμβαίνει στην Ελλάδα για να δω με ποιο τρόπο μας επηρεάζει και εμάς. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες γενικές ερωτήσεις. την περίπτωση της Ελλάδος αφενός αλλά και της Ισπανίας εφετέρου ε, υπάρχουν κάποιες ε, δυνατότητες πίστοσης οι οποίες ε, ως στόχο έχουν να διοχετευτούν κονδύλια στο τραπεζικό σύστημα ώστε να προβλεφθούν κάποιες περιπτώσεις ε, πτώχευσης ή ε, ε, γενικότερης κατάρρευσης της χώρας, ε, τουλάχιστον για την περίπτωση της Ισπανίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν με τις προϋποθέσεις που προκύπτουν τουλάχιστον ε, για την Ισπανία, αλλά όπως εξηγήσατε και εσείς ε, για την περίπτωση της Ελιάδος ε, που ήταν μια περίπτωση γενικότερου προβλήματος, γιατί για μας τα προβλήματα ήταν στον τραπεζικό τομέα κυρίως. Τι δυνατότητες έχουμε σε σχέση με αυτά που έχουμε προβλέψει κάποια στιγμή, δηλαδή πέραν της τραπεζικής εξυγίανσης, η οποία αφορά ένα τμήμα τουλάχιστον της γραμμής προπολογισμού που διατίθεται, αν υπάρχει δυνατότητα δανειοδότησης με συγκεκριμένο στόχο εν τέλει, είτε μέσω τραπεζών είτε μέσω Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που να έχουν όμως ως τελικό στόχο ε, να αποφύγουμε την αποτυχία των, και πτώχευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, να βοηθηθούν οι οικογένειες ε, και ούτω καθεξής. Διότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Οι τράπεζες χρησιμοποιούν τα κονδύλια για να λύσουν τα εσωτερικά τους προβλήματα, δεν ανοίγουν όμως γραμμές δανειοδότησης για τους υπολείπους και επομένως ξεκινά ένας φαύλος κύκλος συνεχούς δανειοδότησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματίες και οικογένειες ε, ε, χρησιμοποιούν τα τελευταία τους ε, χρήματα και αυτό που μπορεί να προκύψει είναι να προκύψει ένας δεύτερος κύκλος μέσω των οποίων οι τράπεζες θα χρηματοδοτούνται και πάλι γιατί δεν υπήρχε ένας τελικός στόχος, ένας τελικός αντικειμενικός σκοπός να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβεβαιώσουν και δημιουργούμε συνεχώς άλλα προβλήματα. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχουν ε, δυνατότητες να είμαστε πιο ευέλικτοι και πιο δημιουργικοί ώστε να δημιουργήσουμε δυνατότητες χρηματοδότησης ε, για να αποφύγουμε αυτό το φαύλο κύκλο της ε, συνεχούς χρηματοδότησης των τραπεζών. Δεύτερον, από ό,τι βλέπω ε, και στην Ελλάδα, όπως έγινε και στην Ισπανία, ξεκινούν μια σειρά από διμερείς πρωτοβουλίες μεταξύ κρατών μελών. για παράδειγμα, στην Ισπανία είχαμε βοήθεια από πλευράς Γερμανίας χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν περνούν από τους κοινοτικού διάβλους. Ε, σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτές οι πρωτοβουλίες που είναι σαφές και ότι οι πολίτες δεν το γνωρίζουν. Οι Ισπανοί ας πούμε ξέρουν ότι υπάρχει μια γραμμή χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που δεν ξέρουν όμως ότι μας τη δίνουν οι Γερμανοί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Ε, θα μπορούσε να υπάρχει ένα πλαίσιο ώστε όλες αυτές οι διμερείς πρωτοβουλίες να εξηγούνται και να υπάρχει και μια σχέση με το τι συμβαίνει από πλευρά Τρόικα. Διότι εμένα μου δίνεται λίγο η εντύπωση ότι ο καθένα κάνει ό,τι του καπνίσει και χωρί να ξέρουμε τι ακριβώ συμβαίνει και γιατί. Το ίδιο και με την εγγύηση για τους νέους, τους οποίους ε, ε, αναφερόμαστε συνεχώς. Λέμε ότι θα έχουμε 40 δισεκατομμύρια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ούτω καθεξής είναι όλες διμερείς πρωτοβουλίες για κάτι το οποίο είναι ακόμα υποσυζήτηση ε, στις πολιετές ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, για το τι θα γίνει και αν θα χρηματοδοτηθούν και θα ήθελα να ξέρω μέχρι ποιου βαθμού υπάρχει μια κάποια ευθυγράμμιση. Αν υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και αν ξέρουμε πού στοχεύουμε. Διότι δεσμεύουμε δημόσιο χρήμα, ευρωπαϊκά κονδύλια και δεν ξέρουμε πού πάνε τελικώς. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτή τη στιγμή, και το είπατε κι εσείς, για την Ελλάδα, επειδή υπάρχει μια απογοήτευση και βλέπουμε ότι οι πόροι τελικώς δεν φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα, οι, οι οικονομικές δομές έχουν ε, ε, καταρρεύσει περισσότερο από ό,τι φανταζόμασταν. Ε, σε ποιο βαθμό λοιπόν υπάρχει ένα αξιόπιστος τελικός στόχος, ε, δηλαδή να μην χάνεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπινων πόρων, υπάρχει κάποια εγγύηση ότι όλα αυτά τα προληπτικά μέτρα ή οι προηγούμενες μελέτες βάσει των οποίων λαμβάνονται μέτρα είναι αξιόπιστα, εγγυώνται κάτι και ότι δεν θα καταρρεύσουν τα πάντα πίσω μας διότι λαμβάνονται κάποιες πρωτοβουλίες και μετά βλέπουμε ότι ούτε θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται και ούτε υπάρχουν δυνατότητες αντίδρασης ούτε τίποτα. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα μέσω των οποίων τα μέτρα για την ανάπτυξη ε, digamos, limitación o, o, ¿cómo decir? Eh, austeridad. Και όλη αυτή η λιτότητα την οποία αποκαλείτε εσείς και επικαλείστε συνεχώς ε, θα μας οδηγήσουν κάπου σε ανάπτυξη, διότι είδαμε ανθρώπινοι πόροι, κοινωνικό ταμείο, όλες αυτές τις παρουσιάσεις πόσο χρόνια δημιουργούν ε, θέσεις εργασίας όλες αυτές οι επενδύσεις που γίνονται. Πού χρησιμοποιούνται όλες αυτές οι θέσεις εργασίας. Αναφερθήκαμε σε μια παγκοσμιοποιημένη ε, αγορά εργασίας, αλλά δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της αγοράς εργασίας, διότι δεν υπάρχουν κοινοί κανόνε. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε λοιπόν εσείς κάποιο χρονικό ορίζοντα. Ξέρετε μέχρι πού πρέπει να επιμείνουμε ώστε να μπορέσουμε να βγούμε ε, νικητές από όλη αυτή τη διαδικασία εφαρμογής μέτρων. διότι θα πρέπει ε, να βρούμε μια λύση ή αλλιώς θα βουλιάξουμε όλοι μαζί και θα προσπαθούμε να επιβιώσουμε και δεν θα ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή την ε, οικονομία που καταβοραθρώνεται ούτε στην Ελλάδα ούτε στις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους και να τους ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσες και επικοδοματικές εισηγήσεις τους. Επίσης καλωσορίζω το έργο της Επιτροπής και της Task Force σε μια περίοδο όπου το Γενικό Κράτος καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την δημοσιονομική εξηγίαση και επίτευξη ανάκαμψης και ανάπτυξης. Η ερώτηση που θέλω να επιβάλλω τόσο στον κύριο Ράχενμπαχ όσο και στον κύριο Πόπεντς είναι η εξή Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε τους κύριους τομείς τους οποίους έχει σημειωθεί η στέρηση και θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Ελλάδα ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων τόσο κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο όσο και κατά την επόμενη. Ευχαριστώ. Thank you very much for such a very clear... Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή αυτή ερώτηση. Κύριε Σόντερκάρτ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σχόλιο για να ξεκινήσω. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι μεγάλη αμηχανία ε, ως προς την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που άκουσα με τόση προσοχή, γιατί μας, λένε, μας λέτε ότι τα πράγματα όλα πάνε πολύ καλά. Προς τη σωστή κατεύθυνση, μας ότι μπήκαν στο σωστό δρόμο. Και έτσι μου ήρθαν ε, στο μυαλό κάποιες δηλώσεις της Τρόικα στην Ελλάδα, για την Ελλάδα που αποδεικνύονται διαρκώς εσφαλμένες. Κάθε φορά η πολιτική που επιβάλλεται φέρνει χειρότερα αποτελέσματα από ό,τι είχαν προβλεφθεί. Έχω λοιπόν αυτό το παράξενο αίσθημα ότι ενώ η Επιτροπή μας λέει ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, ή προ τη σωστή κατεύθυνση, τελικά πάνε προ το χειρότερο. Εν πάση μια ερώτηση για τον κύριο Ράχενμπαχ καταρχά. Σε μια συνέντευξη στη Frankfurter Allgemeine, τη γερμανική εφημερίδα, τη 9η Φεβρουαρίου 2012, ο πρώην Υπουργό των Οικονομικών τη Ελλάδα, ο κύριο Χρυσοχοίδη, είπε, λέει ο μιλητή, είπε ότι οι υψηλές δαπάνες έχουν καταστρέψει την, την ελληνική οικονομία. Αυτή η δήλωση αφορούσε το 2011 και έλεγε ότι τα περιφερειακά ταμεία χρησιμοποιούνται μάλλον για κατανάλωση παρά για ε, επενδύσεις σε μια πιο ανταγωνιστική τεχνολογία και ανάπτυξη. Ερωτώ λοιπόν, αυτές τις κριτικές Τις έχετε λάβει υπόψη, έχουν υπόσταση. Έχετε έρθει σε επαφή κύριε Ράιχενμπαχ με τον πρώην Υπουργό των Οικονομικών, λέει ο μιλητής, ε, για να δείτε τι γνώμη έχει και να το μελετήσετε και να σωματώσετε ενδεχομένω στο έργο της Task Force αυτές τις παρατηρήσεις. Δεύτερη ερώτηση προς τον κύριο Μάνο. Στην ε, παρατήρησή σας σήμερα λέτε ότι έχετε ασχοληθεί με, την, ε, με τις επενδύσεις για το μετρό στην Ελλάδα και τις υποδομές κτλ. Και το αεροδρόμιο. Εδώ ξέρουμε ότι μεγάλο κομμάτι του ελληνικού προϋπολογισμού έχει αφιερωθεί στις υποδομές σε μεγάλο βαθμό οι υψηλέ δαπάνες για όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγάλες, ε, στο μεγάλο έλλειμμα. Η γέφυρα για το Ρίο, οι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, όλα αυτά. Γιατί, ε, και καθώς εδώ έχουμε και συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα θέλω να μου πείτε τι έχετε να πείτε για αυτές τις υψηλές δαπάνες. Οι κατηγορίες είναι αβάσιμες Τα έργα αυτά έχουν υλοποιηθεί κατά τρόπο σωστό, άψογο. Υπάρχουν εμπλοκές με εταιρείε μεγάλες όπως οι Siemens που ανέλαβαν τα έργα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ζικμόντος. Μπαλτσίτης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. του Išvesti susidariusi, iš susidariusi. Δυστυχώ έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα προ το παρόν με τη διερμηνία, θα το λύσουμε αμέσω. Είναι ne tik tais pietietiškos valstybės, bet yra ir šiaurės regione, ir rytų regione. Κύριε Čia ir, ir mano valstybė, kuri irgi taip pat turi didelių problemų dėl taupimo kažkada. Κύριε Πρόεδρε, πολλά άλλα κράτη έχουν ε, δυσκολίες οικονομικές και η δική μου η πατρίδα η οποία αναγκάστηκε να εισαγάγει μια πολύ σκληρή πολιτική λιτότητας Η εφημερία της Ελλάδας έχει στηριχθεί πάνω στην χρηματοδότηση των τραπεζών, στη μεγάλη τραπεζική αυτή ευημερία και τη χρηματοδότηση, τη φούσκα ουσιαστικά, η οποία έσκασε πρώτα βέβαια στις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί βέβαια η οικονομία δεν, έχει, ε, δεν γνωρίζει σύνορα, και ανακαλύψαμε ότι πρέπει να ε, επιστραφούν τα χρήματα αμέσως πρέπει να στηριχθούν οι τράπεζες αμέσως και όχι μακροπρόθεσμα γιατί βρίσκονται σε πολύ δεινή κατάσταση και χρειάστηκαν πολλά χρήματα. Το πρόβλημα το γνωρίζω και, το, γνωρίζω και τις σημαντικές διστάσεις της ανεργίας, αν και δεν έχω να δώσω ε, συνταγές για το πώ μπορεί να δημιουργηθούν θέσει εργασία, αν και με κάποια προγράμματα υποδομών μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες θέσει εργασία. Χωρί όμω να, αυτά να αρκούν. Υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν και στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η η οικονομία η οποία έχει τόσο πολύ εξαρτηθεί από τις ε, εισαγωγέ, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εσωτερικής παραγωγής, θα πρέπει να ε, μεταστραφεί στην ε, βελτίωση της παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο έχουμε και στον, στον κοινωνικό τομέα. Βλέπουμε ότι δισεκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στις κοινωνικές παροχές στην Ελλάδα ή ότι χρειάζονται τεράστια κονδύλια για να υποστηριχθούν οι ανθρώπινοι πόροι. Τι κάνουμε όμως για να βελτιώσουμε στην πραγματικότητα την κατάσταση των ε, πολιτών, για να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες και προσόντα. Στην ουσία τι κάνουμε και βέβαια τι κάνουμε ως προς την μεγάλη πρόκληση που είναι η διοικητική μεταρρύθμιση. Σε αυτή τη μεταρρύθμιση θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μία αποπολιτικοποιημένη χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δηλαδή τα κονδύλια που διατίθενται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να μην βρίσκουν μπροστά τους εμπόδια από αυτούς που είναι ε, ουσιαστικά επιφορτισμένοι με την διάθεσή τους, με την εκτέλεση των προγραμμάτων. Και όπως είπε και η κυρία Γιάλα Σέντερ, πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα και να εξηγήσουμε στους πολίτες και στα κράτη αυτά πόσα πράγματα γίνονται, πόσα ποσά διατίθενται για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, για την μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, για όλα αυτά. Ή διαφορετικά ίσως θα πρέπει να αναστήσουμε άλλα μοντέλα και διαφορετικούς ανθρώπους που θα χειριστούν τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαρτσίτης. Και παρακαλώ τώρα τον κύριο Σκυλακάκη να λάβει το λόγο. Thank you, uh, Mr. President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας όλους τους ε, προσκεκλημένους μας που ήρθαν εδώ να κάνουν τις ε, ομιλίες τους. Και ρωτώ τον κύριο Ράχενμπαχ, αλλά και τους λοιπούς εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Εγώ πιστεύω ότι με καλή πρόθεση προσεγγίζουν όλοι το πρόβλημα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την ουσία των προβλημάτων η Task Force είναι εύστοχος και θα είμαι πιο συγκεκριμένος για να αντιληφθείτε τι εννοώ με την ερώτηση. Τρία είναι τα προβλήματα στον ε, δημόσιο τομέα της Ελλάδας, όλοι το παραδέχονται. Πελατολο... Πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, μεγάλος όγκος του δημόσιου τομέα. Για να δούμε λοιπόν τώρα την πρόσβαση στις, στους σπόρους. 2,9 δις από την ευρωπαϊκή πλευρά έχουν διατεθεί, αλλά μόνο 132 εκατομμύρια ευρώ ε, πήγαν στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα, το ίδιο έτος 2012, γιατί αυτά τα λέει η έκθεση, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα στην Ελλάδα μπόρεσαν να αποσπάσουν από τις τράπεζες 30 επιπλέον εκατομμύρια που εγγράφονται ως ε, δάνεια, ως χρέος δηλαδή, 30 ακόμα εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ουσιαστικά διακρατεί τώρα ο δημόσιο τομέα. Τα δύο κόμματα που εναλλάχθηκαν στην εξουσία. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Δανείστηκαν από τι τράπεζε και αυξάνουν το επίπεδο της χρηματοδότησής τους από το 245 εκατομμύρια στα 270 και εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ικανά, πολύ ικανά τα κόμματα αυτά να διαθέτουν ε, χρήματα ε, στα κόμματα τους, ε, αλλά στο δημόσιο τομέα δεν βλέπω να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν και γι' αυτό θα ήθελα κάποια σχόλια. Για τον δημόσιο τομέα και τις προσλήψεις συζητούμε πώς θα βελτιωθεί ο δημόσιος τομέας κτλ. Αξιοκρατία δεν υπάρχει. Αξιοκρατικές διαδικασίες για τα ανώτερα αξιώματα, τα, τους αξιωματούχους υψηλότερους στον δημόσιο τομέα δεν υπάρχει, όπως έχει παραδεχθεί και ο αρχηγός του δεύτερου σε μέγεθος κόμματος, ο κύριος το δεύτερο κόμμα κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, ε, υπάρχει ένα σύστημα 4-2-1, δηλαδή 4 για το πρώτο κόμμα, 2 για το δεύτερο κόμμα της κυβέρνησης και 1 για το τρίτο κόμμα της κυβέρνησης. Μοιράζονται τις θέσεις, ανώτερες θέσεις στο ε, δημόσιο τομέα. παρέμβαση δε από την Τρόικα ή την Task Force είδαμε μόνο στον τομέα της ε, φορολογίας. Και θα ρωτήσει ο κόσμος, λέει τι θέλετε, θέλετε αξιοκρατία μόνο για την εφορία, όλος ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας δεν χρειάζεται αξιοκρατία για τις ε, θέσεις, τις ανώτατες, ας πούμε, πολιτικές θέσεις στα Υπουργεία κτλ. Και θα προχωρήσω σε ένα πιο συγκεκριμένο ζήτημα. Η κύρια πρόθεση για ιδιωτικοποίηση είναι το ζήτημα των ε, παιχνίων. Το προπό, ο ΠΑΠ δηλαδή. Το στοίχημα και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είστε στενήμεροι για όλα αυτά. Ξέρουμε πάντως ότι γίνεται πολύ μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσα από αυτό το στοίχημα. Όλα αυτά τα χρόνια, 5-6 χρόνια, έχουμε μεγάλα σκάνδαλα εγκληματιών που συνελήφθησαν να νομιμοποιούν παράνομα έσοδα μέσω αυτού του συστήματος των στοιχημάτων και των λαχνών του ΟΠΑΠ, είτε πρόκειτο για ναρκωτικά, είτε πρόκειτο για δίκτυα πορνείας, είτε πρόκειτο για γεωργιανή και ρωσική μαφία, είτε πρόκειτο για ε, φοροφυγάδες γιατρούς και δικηγόρους, είτε πρόκειτο για ε, διεφθαρμένους εφοριακούς, όλοι νομιμοποιούν μέσω του ΟΠΑΠ τα έσοδά τους. Έτσι λοιπόν ο ΟΠΑΠ από δημόσιο μονοπόλιο στο οποίο εμφανίζονται τα σκάνδαλα αυτά μετατρέπεται σε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο χάρη στην ιδιωτικοποίηση. Έχετε ποτέ ασχοληθεί με το πρόβλημα της νομοποίησης παράνομου χρήματος εκεί. Και κοιτώντας την έκθεση της Task Force που μας λέει ότι έχει δώσει τέσσερα σεμινάρια με επίπεδο ε, ευαισθητοποίησης Α1 για, το, ε, παράνομο, για την ομοποίηση παράνομου χρήματος και το ξέπλυμα χρήματος. Κοιτάξτε να σας πω, ευαισθητοποίηση υπάρχει, δεν υπάρχει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Πρέπει ουσιαστικά δράση να αναλυφθεί στους συγκεκριμένους αυτούς τομείς μέχρι να αλλάξει κάτι. Και θα συνεχίσω με κάτι ακόμη για να ολοκληρώσω εφοριακή και διαφάνεια. Στην τελευταία έκθεση της ε, Διεθνούς Διαφάνειας, Transparency International, για την Ελλάδα, για το σύστημα της συλλογής φόρων στην Ελλάδα, καταγράφεται ότι με βάση τις απαντήσεις στις δημοσκοπήσεις ο πολίτης έχει δώσει τουλάχιστον 80.000 φορές φακελάκι σε εφοριακούς, μόνο σε εφοριακούς. 80.000 μέσα στο έτος 2011, 12. Αν λοιπόν μετρήσουμε πώς είναι η εφοριακή, ε, κάθε τρεις εργάσιμες μέρες ένας εφοριακός παίρνει φακελάκι. Δωροδοκείται. Ερωτώ λοιπόν τι κάνετε γι' αυτό. Έχετε περιγράψει μια στρατηγική ειδική για την καταπολέμηση της διαφθοράς, έχετε εισαγάγει προτάσεις για τη διοντολογία των δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Ερωτώ, έχει κάνει κάτι το ουσιαστικό η Task Force έχει στοχευμένη δράση. Είμαι πεπισμένος για τις καλές της προθέσεις. Είμαι πεπισμένος ότι κάνει όλα αυτά τα ωραία τα σεμινάρια, ότι κάνει αυτές τις στρατηγικές, καταρτίζει ιδέες και ε, προγράμματα. Αλλά κάνετε κάτι το οποίο να φέρνει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντικές και γενικές ερωτήσεις. Ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον Στέφανο Μανοπίου με μεγάλη ευτυχία. Μίλησε για την Ιερή Αγελάδα, το δημόσιο τομέα δηλαδή στην Ελλάδα και είπε ότι ό,τι πέτυχε μέχρι τώρα η Τρόικα το πέτυχε μέσω του εκβιασμού. Δηλαδή, αν δεν κάνετε αυτό που σας λέμε, δεν θα πάρετε τα χρήματα που σας έχουμε υποσχεθεί. Είναι ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί κάποια αλλαγή ή, αν θέλετε, αφελής προσέγγιση του ότι δεν αρκεί να συμβουλεύει, να προτείνει κανείς, αλλά πρέπει να το κάνει, όπως είπε ο κύριος Μάνος εξάλλου, ίσως θα πρέπει να αλλάξει λίγο την προσέγγιση. Μήπως από την αρχή ήσασταν λίγο πολύ αφελής; Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, προσέγγισή σας όσον αφορά τα διάφορα ποσοστά που μα παρουσιάσετε για την Ελλάδα και Κύριε Πόμπερ, μιλήσατε για τα ποσοστά χρηματοδότησης και απορρόφησης των κονδυλίων. Δώσατε στοιχεία για το 12 και το 13 λέγοντας ότι 11 δισεκατομμύρια έχουν εκταμιευθεί και περίπου 7 έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν πληρωθεί. Εκρεμούν. Δεν έχουν εν πάση περιπτώσει, δοθεί, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για σχέδια της πραγματικής οικονομίας, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών των κονδυλίων που μπαίνουν σε αυτά τα επίπεδα απορρόφησης, ουσιαστικά έχουν εγκριθεί, τελικά όμως δεν έχουν εκταμιευθεί, δεν έχουν δοθεί. κύριε Ράχιμπακ, κύριε στον κατάλογο των ε, διαφόρων ε, προγραμμάτων και σχεδίων στα οποία εμπλέκεστε και τα οποία είναι προγράμματα προτεραιότητας όπως τα αποκαλείτε, πάνω από 160 προγράμματα. Αναφέρεστε σε σχέδια του 2011. Μα δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Κύριε Στούμπ, αναφερθήκατε στην προσαρμογή της προσέγγισής σας, της πολιτικής σας, της μεθόδου που χρησιμοποιείτε και σας πιστεύω όταν το λέτε. Κάνω λοιπόν την εξή ερώτηση. Πόσες θέσεις απασχόλησης δημιούργησε το χρηματοδοτικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα σύστημα στην Ιταλία, στην Σικελία, που χρησιμοποιεί τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά και την ίδια ώρα τα κονδύλια που έρχονται από τα κοινωνικά ταμεία για την δημιουργία συγκεκριμένων ε, επιχειρήσεων. Ο, η νομοθεσία στην Ελλάδα το προβλέπει. Έχετε δει όμως να έχουν δημιουργηθεί τέτοιες επιχειρήσεις ελάχιστες στην Αθήνα και ε, κάποιες στην ΚΟ. Γιατί, δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά γιατί εκεί υπάρχει ένας πολύ δραστήριος δήμαρχος, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια κρίσης, δεν έχουν δημιουργηθεί θέσεις απασχόλησης σε αυτό το τομέα, μετά από τη χρηματοδότηση και την ε, πρόσβαση στα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Ταμείων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παραδείγματο χάρη. Κύριε Κνάπεν, τελευταία μου ερώτηση είναι για εσά. Σα ευχαριστώ πολύ γιατί μα δώσατε πολύ σημαντικά στοιχεία, αριθμού, τι κάνετε, συγχαρητήρια. Γιατί όντω έχουν υπογραφεί πολλέ συμβάσει. Αναφερθήκατε σε μια πολύ συγκεκριμένη σύμβαση που είναι το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Και λέτε ότι θα απορροφηθούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ η ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ ε, ευφυής και χρησιμοποιεί καινοτομία. Το θέμα όμως είναι ότι σήμερα τα μεγάλα τέτοιου είδους σχέδια δεν μπορούν πλέον να αποφέρουν ωφέλη. Τελείωσαν τα μεγάλα προγράμματα και σχέδια. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ταμείο Εγγύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και είχε αρχικά προβλεφθεί το ξεκίνημα της λειτουργίας του το Μάιο. Πότε επιτέλους θα ξεκινήσει όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλοι συμφωνούμε εδώ, όλα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, ότι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης είναι μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λείπει όμως εδώ η χρηματοδότηση. Γιατί, σας ερωτώ, φταίει η ελληνική κυβέρνηση, φταίει η Τρόικα, γιατί δεν βρίσκει τρόπο μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και μέσω των μηχανισμών παρέμβασης δεν βρίσκει τρόπο να κινητοποιήσει αυτό το μηχανισμό. Ευχαριστώ πολύ ο Ζαν Πολοντίνο, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι τρομακτικά αυτά που ακούω σήμερα εδώ. Έχω την εντύπωση ότι όταν στις εκλογές θα αρχίσουμε να μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Εγώ συγχαίρω τους υπαλλήλου της Επιτροπής, την Τρόικα, για την υπομονή τους, την επιμονή τους. Δεν είναι εύκολη κατάσταση στην Ελλάδα με αλλαγή κυβερνήσεων, με αντιστάσεις, να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν τέτοιες δύσκολες αποφάσεις θα κάνω τρεις-τέσσερι παρατηρήσεις. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες. Ξέρουμε σήμερα αν έχουν ενημερωθεί σωστά οι Έλληνες πολίτες. Τι έγινε στο παρελθόν, τι έγινε με τα κοινοτικά κονδύλια. Και εγώ πολλές φορές διαβάζω στον τύπο ότι οι Έλληνες λένε εμείς δεν ξέρουμε γιατί χρήματα πρόκειται, δεν ξέρουμε από πού προέρχονται, και γιατί πρέπει εμείς να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα. Μα πρέπει να τους ενημερώσουμε. Και θα πρέπει να υπάρξει ευαισθητοποίηση αυτών που τους εκπροσωπούν των ε, Ελλήνων βουλευτών. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι η ευθύνη των τραπεζών. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ε, επικρίνουμε περισσότερο τις τράπεζες. Κάθε φορά που μια τράπεζα δανείζει σε ένα υπερχρεωμένο φορέα, Σφάλι. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα είναι ότι δόθηκαν υπερβολικά πολλά κονδύλια, δάνεια στη χώρα αυτή. Ξέρω βεβαίω ότι σήμερα το ποσό αυτό έχει μειωθεί στο 50%, αλλά αυτό ίσως δεν αρκεί. Και όταν βλέπω τι έγινε στην Κύπρο, ο ερασιτεχνισμός φαίνεται να έχει επικρατήσει και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε διδαχθεί το μάθημα της Ελλάδας. Αυτό διαπιστώνω. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω πραγματικά πως λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί το Συμβούλιο, η Επιτροπή και ελπίζω όχι και η Κεντρική Τράπεζα δεν ακολουθούν τις επιθυμίες της Επιτροπής μας όσον αφορά την επιτήρηση Τόσα χρόνια ζητάμε μια εποπτεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων. Και για να διατηρήσει αυτή η τράπεζα το τριπλό αλφα της, θα πρέπει πραγματικά να υπάρξει μια τέτοια εποπτεία. Θα ψηφίσουμε την Τραπεζική Ένωση και θα έχει παραμείνει το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του ελέγχου και της εποπτείας της έκρεμες. Πρόεδρος. Καταλαβαίνω ότι θα πάρετε το λόγο για να απαντήσετε τις ερωτήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω τα εξή συνοψίζοντα. Όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια καλή θέληση από μέρου του Τρόικα. Όλοι συμφωνούν ότι γίνονται προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες. Καλή θέληση λοιπόν και προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Επενδύσεις σε έργα υποδομής, δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων. Επενδύσεις που αντιμετώπισαν προβλήματα στο παρελθόν. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες και για να φτάσει σε μια βιώσιμη ανάκαμψη που θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη. Γιατί μέχρι τώρα επιγόντως χρηματοδοτούμε κάποιους τομείς. Το δίλημα λοιπόν είναι Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια αηφόρο ανάπτυξη. Και θα δώσω αμέσως το λόγο στους ομιλητές, τον κύριο Ράιχενμπακ, τον κύριο Μάνο, Όπενς, του και Κνόπεν. Εντάξει. Κύριε Ράιχενμπακ, είστε ο πρώτος ομιλητής. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πόπεν θα πρέπει να φύγει από ό,τι μου είπε. Αν δεν σας πειράζει λοιπόν να αλλάξουμε λίγο τη σειρά, να απαντήσει πρώτος, γιατί εγώ θα παραμείνω τους ή άλλους. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Ε, θα μείνει όμως ο συνάδελφος, ο ειδικό για το ελληνικό τμήμα, αλλά εγώ δυστυχώς πρέπει να φύγω. Θα ήθελα να σταθώ στις βασικές προκλήσεις καταρχάς. Όπως σας είπα και στην παρουσίασή μου, αναλύσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα από πλευράς εφαρμογής των κονδυλίων, αλλά κοιτάξαμε και ευρύτερα ποιες είναι οι προκλήσεις. Και φυσικά οι βασικές προκλήσεις είναι το γεγονός ότι το οικονομικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο και δεν είναι ανταγωνιστικό. Και αυτό φυσικά θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα για τα ταμεία και σχετίζεται και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις καινοτομίε, την έρευνα και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό ακριβώ και θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ιδίω αν το συγκρίνουμε σε χρηματοδότηση υποδομών. Ε, δεν μπορούμε να λέμε ε, ότι αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Ε, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέτρων. Ε, κέντρα ανάπτυξη για τι επιχειρήσει, για παράδειγμα και να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή υποστήριξη την οποία θα πρέπει να δημιουργήσουμε και όλα αυτά θα πρέπει ε, να προχωρήσουν και να προχωρήσουν και τα διευρωπαϊκά δίκτυα και έχουμε μεγάλο προβληματισμό όταν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ε, τοπικά οδικά δίκτυα και το καθεξής. Ε, θέλουμε να έχουμε λοιπόν ένα καλό ρυθμιστικό πλαίσιο και αυτό νομίζω ότι είναι και η απάντηση για όλους. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν είναι τα συνήθεια είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο και αν το συγκρίνουμε με την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο είναι ένα τελείως καινούριο ε, πλαίσιο το οποίο δίνει περισσότερες δυνατότητες να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα, να προσανατολιστούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό είναι λοιπόν το οποίο θέλουμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε με τα κράτη-μέλη και με τις ελληνικές αρχές εν γέννη. Χρειαζόμαστε πλήρη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, διότι τα προγράμματα τα οποία θα γίνουν εκεί στις περιφέρειες ε, θα είναι επιμερισμένες διαχείρισης. Και γι' αυτό ακριβώς μία από τις προκλήσεις είναι να αντιμετωπίσουμε αυτή την αναεπαρκή δημόσια διοίκηση που όπως λέμε και στο έγγραφό μας ε, αποτελεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση για το επόμενο ε, διάστημα για να ενισχύσουμε τη δημόσια διοίκηση και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα τις συμβάσεις και το τι έχει γίνει με τη χρηματοδότηση. Έχουμε πληρώσει το 54% των συμβάσεων. Αλλά αν δείτε επιτόπου τι γίνεται, έχουμε εγκεκριμένες συμβάσεις της τάξης του 85% και αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου ε, μία υπερβολική σύναψη συναβάσεων επιτόπου, εκκρεμεί ένα 30%. Αυτό είναι θετικό μεν γιατί σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση για τα κονδύλια αυτά, αλλά αν κάνετε τη σύγκριση στα στοιχεία υφέρπουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι αδρανή προγράμματα, γι' αυτό και ακριβώ αναφέρθηκα και στην κατάλληλη οριμότητα των προγραμμάτων, γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα στην Ελλάδα. Υπάρχουν έργα τα οποία αποφασίζονται και κατόπιν ε, δεν είναι σαφή ποιος είναι ο κύριος του έργου και τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν. Προσπαθούμε να έχουμε ένα κατάλογο ε, των βασικών προγραμμάτων. Αυτός ε, δημιουργήθηκε, έχουμε αυτά τα 181 προγράμματα και το βασικό στοιχείο λοιπόν είναι να έχουμε ως όριο το 2015, γιατί μέχρι τότε πρέπει να έχουν περατωθεί αυτά τα έργα και τα ημιτελή έργα μπορεί να αποτελέσουν τεράστιο πρόβλημα και να οδηγήσουν σε δημοσιονομικές διορθώσεις, γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι επειδή έχουμε χρόνο πρέπει να το επεξεργαστούμε. Έχουμε μια αργή πρόοδο, αλλά όπως το θέμα των συμβάσεων παραχώρησης για τα οδικά δίκτυα, είναι πολύ αργή διαδικασία και πρέπει κάπως να την ολοκληρώσουμε. Είμαστε όμως αισιόδοξοι διότι θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του 2015 μπορούμε να προχωρήσουμε και να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Αυτό ήθελα να πω και ζητώ συγγνώμη που πρέπει να φύγω, αλλά θα μείνουν οι συνάδελφοι εδώ για να απαντήσουν τυχόν ε, περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράχεμπαχ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες αυτές τις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πρώτη παρατήρηση. Αν κοιτάξουμε τι συνέβαινε πριν από ένα χρόνο και συγκρίνουμε, θα θυμούνται ίσως οι περισσότεροι εδώ την κατάσταση πριν από ένα χρόνο που ο μεγαλύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους. Μιλούσε για την πιθανότητα του Brexit της Ελλάδας, της εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Κατά 90% πιθανολογούνταν αυτή η έξοδος. Τώρα δεν νομίζω να πλησίαζε κανείς στις προβλέψεις του τέτοιου είδους ποσοστά. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή. Και μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση έχει αντικειμενικά βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε ύφεση, αλλά υπάρχουν σαφή μηνύματα ότι θα παρουσιάσει επιδόσεις ρεκόρ ο τουρισμός εφέτος, ότι θα έχουμε ε, σημαντική άνοδο στις εξαγωγές εφέτος, ότι αρκετοί οικονομικοί δείκτες εφέτος παρουσιάζουν κάποιες έστω ελαφρές βελτιώσεις. Ύστερα από μήνες, πολλούς μήνες αύξησης της ανεργίας φαίνεται να αλλάζει η κατάσταση και να αντιστρέφεται ο λόγος των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε σχέση με αυτές που χάνονται. Και άρα υπάρχει από ό,τι φαίνεται ένα δυναμικό, μια δυνατότητα για βελτίωση, για ανόρθωση της κατάστασης στην Ελλάδα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν να δούμε σε ποια σημεία η Ελλάδα μπορεί και στο μέλλον να σταθεί και να βελτιώσει ακόμη τη θέση της. Ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό περιβάλλον, στις αδειοδοτήσεις, στις προμήθειες, στη μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις ε, άμεσες επενδύσεις, για τις ξένες επενδύσεις, για να φέρουν αποτέλεσμα και να είναι ε, αποτελεσματικές. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτό που εμείς προσφέρουμε μαζί με πολλούς διεθνείς οργανισμούς, τον ΩΣΑ, την Παγκοσμία Τράπεζα και άλλους, ως συμβουλές και να τις υλοποιήσει κατά τρόπο αποφασιστικό, κατά τρόπο καταχή, ώστε να αποκατασταθεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Και επίσης, το τεράστιο πρόβλημα που αναφέρατε όλοι σας, το πρόβλημα της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία έχει ξεπεραστεί. Οι τράπεζες θα βρεθούν ακόμη σε δύσκολη κατάσταση, όπως πολύ σαφώς περιέγραψε ο κύριος Μάνος, για κάποιους μήνες ή και χρόνια ακόμη. Αλλά μπορούν σε αυτό τα διαρθρωτικά ταμεία να δώσουν μια βοήθεια, μαζί βέβαια με τη δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την και από, άλλους πηγές, και από άλλες πηγές και διμερείς ακόμη που έχουν αναφερθεί. Όμως, η συνειδητοποίηση του ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και του ότι χρειάζονται για να το ξεπεράσουμε συγκεκριμένα μέτρα έχει ουσιαδέστατη σημασία. Έχει γίνει προπαρασκευαστικό έργο για τη δημιουργία ε, των υποδομών για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Έχει ήδη δοθεί το περίγραμμα αυτών των μεταρρυθμίσεων και πλέον πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει τα απαραίτητα βήματα ώστε να υλοποιήσει αυτά τα έργα. Και για να απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση της κυρίας Αγιάρα Σέντερ, Υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά με το χρηματοπιστωτικό σύστημα Υπάρχουν κράτη-μέλη που με ανακεφαλαίωση των τραπεζών τους παράλληλα έχουν περιγράψει ενδείξεις, κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες, να δεσμευθούν τουλάχιστον ηθικά, αν όχι νομικά, να ακολουθούν προκειμένου να υπηρετήσουν την πραγματική οικονομία. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει στην Ελλάδα, δεν έγινε αλλά θα μπορούσε να γίνει ή μη άλλο σε άλλα Ένα άλλο ζήτημα, ερώτημα που ετέθησε σε φως, που, είναι, που εντοπίζονται οι κύριες αδυναμίες. Αναμφίβολα, στο δημόσιο τομέα, στο πρόβλημα, στις αδυναμίες που έρχονται στο σύστημα των εφοριών, ιδιαίτερος, στο θέμα της διαχείρισης των διαθροτικών ταμείων, όπου εντοπίστηκε πως υπάρχει μεγάλο περιθώριο για οι προσπάθειες λοιπόν στις οποίες αποδίονται οι πάντες μαζί με τα διευθυντικά ταμεία, Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, Γενική Διεύθυνση για τα Περιφερειακά και τη δική μας την ομάδα για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και τους προσεχείς μήνες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και βέβαια καταγράφω και, τις, ε, και την παρατήρηση ότι εφόσον θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στη διαχείριση των ταμείων και να προσφέρουμε αρρωγή ουσιαστική πρέπει και αυτό να το πράξουμε λαμβανωμένων υπόψη των δυνατοτήτων στην κάθε περιοχή και των αναγκών και δυνατοτήτων και των δήμων. Ο κύριος Σόντεργκαρτ Αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κύριου Χρυσοχοίδη, πρώην Υπουργού της Αναπτύξεως. Δυσκολεύομαι να απαντήσω στις παρατηρήσεις αυτές, στο ερώτημα του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε εργαστεί χέρι-χέρι προκειμένου να βελτιώσουμε την κατάσταση ως προς τα διορθωτικά τομέα. Και σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες κάποιες βελτιώσεις. Την ομάδα εργασίας άλλωστε, για το περίγραμμα αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ως προς το πλαίσιο για την ανάπτυξη, ήταν ο κ. Σοφιχοίδης που το έφτιαξε. το ερώτημα εάν είναι εύστοχη, εάν έχει αποτέλεσμα η παρουσία μας και το έργο μας. Πρόκειται για μια ερώτηση που απασχολεί οποιονδήποτε να λαμβάνει τέτοιο έργο. Και γνωρίζω βεβαίως ότι υπάρχουν προβλήματα στους τομείς που αναφέρατε, αναμφίβολα. Το ερώτημα είναι, και η απάντηση μαζί. Μπορούν οι ελληνικές αρχές στους τομείς αυτούς να κάνουν τις τομές εποφελούμενες και της προσφοράς βοήθειας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνών Οργανισμού για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Μέσα στον πρώτο χρόνο της ε, ύπαρξης της τρέχουσα κυβέρνηση έχει κάνει πολλά, το είπα και από την αρχή πολλές ακόμη διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να υλοποιηθούν και η τελική κρίση για αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές θα προκύψει ανάλογα με το αν μέσα σε ένα χρόνο δούμε αλλαγές στις δομές, στις διαρθρώσεις και όχι μόνο στην οικονομική κατάσταση. Μεσοπρόθεσμα δηλαδή και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας. Και για αυτήν χρειάζεται να αλλάξουν οι δομές και όχι μόνο να αυξάνονται οι φόροι ή να μειώνονται οι δαπάνες. Και τέλει, θα ήθελα να πω ότι ύστερα από 20 μήνες εργασίας στην Ελλάδα, μαζί με πολλούς Έλληνες και ξένους ε, Ευρωπαίους συναδέλφους γιατί λοιπόν ύστερα από αυτούς τους 20 μήνες γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες και αδυναμίες. Πιστεύω ότι η προσπάθεια στην οποία έχουμε αποδηθεί μαζί με τα κράτη-μέλη για να υποστηρίξουμε την Ελλάδα σε αυτό το τιτάνιο έργο της αλλαγής της δημόσιας διοίκησης, μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, παρουσιάζει κάποια αποτελέσματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας η κυβέρνηση, η τωρινή, έχει δημιουργήσει το θεσμό ενός Γενικού Γραμματέα Συντονισμού. Και αν διαβάσετε την έκθεση, στις αρχές του 2012 αν δεν απατώμε, ήταν που ζητούσαμε τον συντονισμό. Λέγαμε ότι η απουσία συντονισμού ήταν ένα από τα κύρια προβλήματα, μια από τις κύριες δυσλειτουργίες στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπαμε εμείς καθημερινά στη δουλειά μας. Έτσι. Η δυνατότητα με αυτή την θέση του Γενικού Γραμματέα και το συντονισμό υφίσταται, πρέπει τώρα να αξιοποιηθεί και να φέρει αποτέλεσμα, να ε, φυσικά η θέση αυτή, γιατί δεν υπάρχει όλο το προσωπικό, αλλά ε, μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και αναφέρατε επίσης και το πρόβλημα της διαφθοράς. Τουλάχιστον, θα σας απαντήσω, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας έχει περάσει νόμος που επιτρέπει, δίνει βάση για να ε, αναλυφθεί αποφασιστική και ουσιαστική δράση για την πάταξη τη διαφθορά. Μπορεί να έχετε τι επιφυλάξει σα, το αντιλαμβάνομαι σε έναν βαθμό, μπορεί να τι συμμερίζομαι και εγώ αυτέ τι επιφυλάξει, αλλά υπάρχει η νομική πλέον βάση και αυτό είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράιχενμπαχ. Επτά λεπτά έχουμε ακόμα πριν ξεκινήσει το επόμενο τμήμα της συζήτησης και υπάρχουν ακόμα τρία άτομα τα οποία θα πρέπει να απαντήσουν. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχάς τον κύριο Στέφανο Μάνο αν θέλει να απαντήσει σε ερωτήσεις που τα Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω μία ερώτηση άκουσα να μου απευθύνεται. Με την άδειά σα λοιπόν θα δημιουργήσω κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν μου ετέθησαν και θα απαντήσω σε αυτές αν μου επιτρέπετε. Uh, Ετέθη μία ερώτηση για το κατά πόσον η Task Force έχει λόγο ύπαρξης να σας πω το εξής. Αν εγώ ήμουν στη θέση του Σαμαρά, ο κύριος ε, Ράχενμπαχ θα είχε πολύ σημαντικό λόγο ύπαρξης και θα ήξερα πώς να τον χρησιμοποιήσω. Δεν τίθεται θέμα του κατά πόσον ε, χρειαζόμαστε την Task Force, αλλά ε, κατά πόσον το ε, κράτος το οποίο δέχεται τη βοήθεια είναι διατεθειμένο να αλλάξει. Το ερώτημα λοιπόν δεν θα πρέπει να απευθύνεται στην Task Force αλλά στους Έλληνες. Θέλετε να σας βοηθήσει ο Ράιχενμπαχ. Και εδώ έγκυται το πρόβλημα. Και όπως είπα και προηγουμένως δεν είναι σαφές. Ε, αν κατάλαβα καλά, με ρωτήσατε αν θα πρέπει να δώσουμε στους Έλληνες ψάρια ή να τους μάθουμε πώς να ψαρεύουν. Αυτό είπατε κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Εγώ θα απαντούσα σίγουρα να τους διδάξετε πώς να ψαρεύουν. οποιοσδήποτε σόφρον άνθρωπος αυτό θα έλεγε. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι εκπνέουν όμως οι προθεσμίες. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να μάθουμε στους Έλληνες πώς να ψαρεύουν. Επομένως, θα πρέπει να δράσουμε έως και ριζοσπαστικά σε κάποιες περιπτώσεις. Και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να αναφέρω και αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άκουσα με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Κνάπεν να επισημαίνει ότι θα πρέπει να εμείνουμε στην βαθμολογία των τριών α και όχι να μην ε, δεχόμαστε οποιαδήποτε πολιτική πίεση. Εγώ δεν ε, είμαι τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα των εγγυήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί δεν είναι πάρα πολλές οι δομές που θα μπορέσουν να απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Ε, υπάρχουν άλλα άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η χρηματοδότηση των χαμηλότερων μισθών. Σε πολλές τομείς τα πράγματα είναι χαόδη. Και θα ήθελα να πω ε, κάτι το οποίο νομίζω ότι ο κύριος Ράιχενμπαχ ανέφερε από αυτά που είπα προηγουμένως. Πρέπει να υπάρχει μια αυστηρή αναθεώρηση ποιότητας των εισοδημάτων των τραπεζών, των, ε, ε του ενεργητικού τους θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαφάνεια για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να μην επιτρέψουμε να μας ξεφύγει ο έλεγχος όπως ε, συνέβη σε πάρα πολλές περιπτώσεις του κόσμου και ε, προσφάτως και στην Κύπρο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια πολύ στενή εποπτεία της κατάστασης του χρηματοοικονομικού συστήματος και να μην ζούμε σε έναν αισιόδοξο ε, κόσμο ο οποίος όμως δεν έχει γερά θεμέλια. Η ερώτηση που μου ετέθη νομίζω ότι ήταν από τον κύριο Σόντεγκαρτ για τα προγράμματα υποδομών τα οποία ξεκίνησαν όταν ήμουν εγώ υπουργό σου πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 25 χρόνια λοιπόν εγώ τι έκανα. Εισήγαγα την έννοια στην Ελλάδα ότι για κάποια μεγάλα έργα υποδομών καλό θα ήταν αντί να αναλαμβάνει το βάρος ο φορολογούμενος να χρησιμοποιούνται κονδύλια από το χρήστη. Ο χρήστης να πληρώνει το βάρος. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε και ο μειοδετικός διαγωνισμός για το αεροδρόμιο της Αθήνας ε, και ε, εκεί οποιοδήποτε κάνει την προσπάθεια θα ανταμείβεται στη συνέχεια. Το ίδιο έγινε και για τα μεγάλα οδικά δίκτυα. Ε, στο δυτικό τμήμα της Ελλάδος αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι εξωφρενικά. Και αν μπορώ να ε, πω κάτι, θεωρώ ότι οποιαδήποτε επίκριση είναι αβάσιμη. Αν θα μπορούσατε να επικρίνετε το οτιδήποτε, από τότε που είχαμε τα τρία μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα, τίποτα δεν έχει συμβεί μέχρι προσφάτως. Και μόνο το γεγονός ότι το μόνο αεροδρόμιο στην Ελλάδα το οποίο το πληρώνουν οι επιβάτες και όχι οι φορολογούμενοι είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι εξωφρενικό. Κάθε αεροδρόμιο στην Ελλάδα θα έπλεπε πλέον να χρηματοδοτείται από τους χρήστες και όχι από τους φορολογουμένους. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και πάλι για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως στην παρουσίασή μου. Ότι δεν θέλει κανείς να αγγίξει την Ιερή Ελλάδα. Ακόμα και για τα αεροδρόμια. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το αεροδρόμιο γιατί δεν θέλουν να αγγίξουν τους εργαζομένους του αεροδρομίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι αποτελούν απόδειξη ε, στην Ελλάδα και πρότυπο καλών έργων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάνο. Κύριε Κνάπεν, σας δίνω το λόγο γιατί νομίζω ότι πρέπει να φύγετε λίγο νωρίτερα. Ευχαριστώ πρόεδρε. θα απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις που μου απέφθηνε κυρίως ο εισηγητής, ο κύριος Χατζημαρκάκης. Ρωτήσατε για το Ταμείο Κίσων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξεκίνησε. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο. Σταδιακά, αλλά ξεκίνησε. Όπως είπε ο κύριος Δράχενμπακ, όντως το θέμα είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί για τις τράπεζες. Η επισφαλής κατάσταση των ε, τραπεζών. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει, όπως ξέρετε, διπλό θέμα. Και βεβαίως σε αυτό προστίθεται το θέμα της αβεβαιότητας όσον αφορά τις τράπεζες και το θέμα της ε, αξιοπιστίας της πιστοληπτικής ικανότητας, αλλά και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι εμείς δεν είμαστε μία τράπεζα για το ευρύ κοινό. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να περάσουν τα κονδύλια από εμάς τις ελληνικές τράπεζες. Εμείς εγγυόμαστε τα δάνεια που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες. Και βεβαίως υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχουν ε, κανονισμοί και ρυθμίσεις που διέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία. Αλλά όπως είπαμε προηγουμένως προσπαθούμε να αντιδράσουμε, να προσαρμοστούμε στην κατάσταση της Ελλάδας χρησιμοποιώντας εργαλεία του παρόντος και του παρελθόντος. Είναι όμως ευχάριστο και το επαναλαμβάνω ότι ξεκίνησε το Ταμείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε συνεισφέρει με πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα μεγάλα σχέδια στα οποία αναφερθήκατε, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε και έχουμε σχεδιάσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δοθεί έμφαση τις επενδύσεις μέχρι το 2020 σε βιωσιμότητα, σε καινοτομία και όχι μόνο στα παραδοσιακά έργα υποδομής, δηλαδή γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι και σιδηρόδρομοι. Υπάρχουν 181 μεγάλα σχέδια, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση που έχετε τα οποία έχουν κριθεί σαν σκόπιμα, σαν βιώσιμα και σαν προγράμματα που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας. Το μετρό είναι ένα από αυτά. Έχουμε προχωρήσει σε μια μελέτη σκοπιμότητας κόστους ωφέλειας από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες Βεβαίω και θα συνεχίσουμε λοιπόν τέτοιου είδου επενδύσεις. Αλλά φυσικά και στοχεύουμε επενδύσεις ε, στην καινοτομία και στο μέλλον. Κύριε Οντή, μιλήσατε για την, ε, τον έλεγχο της τράπεζάς μας, την ε, επιτήρηση, την εποπτεία. Έχουμε, όπως ξέρετε, το λογιστικό μας συμβούλιο, Audit Committee, την Επιτροπή Εποπτείας. Έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που ελέγχουν τη δράση μας και επίσης αναφερόμαστε σε εσά. Με διαφάνεια. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην ετήσια έκθεσή μας. Σαν παράρτημα της ετήσιας έκθεσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και είμαστε υπόλογοι και υπάρχει διαφάνεια στη δράση μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Κνάπεν, για τις απαντήσεις σας. Ένα τελευταίο σχόλιο, Ζων Πιέροντι. Κύριε Γενική Διευθυντή, δεν μίλησα για τη διαφάνεια. Δεν είπα ότι δεν είστε διαφανείς. Είπα ότι δεν υπάρχει τραπεζική εποπτεία όταν ο Επίτροπος Μπαρνιέ, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, μας λένε ότι όλα τα ιδρύματα θα υπόκεινται σε τραπεζική εποπτεία, εσείς δεν υπόκεινται. Και πραγματικά αυτό που αναφέρετε εδώ, ότι έχετε διοικητικό συμβούλιο κτλ, δεν αρκεί. Λυπούμε που ακούω αυτή την απάντηση. Υπήρχε η πρόταση Τρισέ. Ε. Υπάρχει η τροπολογία που έχω υποβάλει και επαναλαμβάνω μια διαπίστωση. Φυσικά και είστε διαφανείς, αλλά δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Δεν υπάρχει τραπεζική εποπτεία. Κύριε Κνάπεν, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Ναι, απλώς θα επαναλάβω. Κύριε Οντή, συμφωνώ μαζί σας. Δεν αναφερόμαστε σε διαφάνεια, άρα δεν θα επαναλάβω το ίδιο. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βόλφ, ο οποίος είναι ο τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ τον κύριο Κνάπεν. και μπορούμε να συνεχίσουμε. care for Yeah, I now would like to welcome here Guntram Wolf. Καλώς ορίζω εδώ τον Guntram Wolf. Διευθύνοντα του Think Tank Brücker των Βρυξελών. Από ό,τι έχω μάθει ήταν πολλά αυτά τα οποία καταγράψατε από τη σημερινή συζήτηση. Για να δούμε λοιπόν από τις συστάσεις τι μπορούμε να αποκομίσουμε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι θέλω να διατυπώσω συμπεράσματα από το σημερινό ε, από τη σημερινή συζήτηση που ήταν πολύ πλούσια σε παρατηρήσεις. Απλώς θα ήθελα να αναφερθώ σε μια αξιολόγηση για την ε, υποστήριξη προς χώρες της Ευρωζώνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Εθνικό Ταμείο, προγράμματα χρηματοδότηση δηλαδή για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Και αυτές οι παρατηρήσεις βέβαια έχουν ε, και την οικονομική ασφαλώς επισκόπηση αλλά και την θεσμική δομή, δηλαδή την Τρόικα θα επικεντρωθώ, μια και το θέμα μας είναι η Ελλάδα, μόνο στο κομμάτι που αφορά την Ελλάδα, της εκθέσεως αυτής, αλλά εάν μου το επιτρέψει ο χρόνος, στο τέλος θα διατυπώσω συμπεράσματα και για την Τρόικα. Ως προς την σύγκριση μεταξύ των τριών κρατών το πρόγραμμα για την Ελλάδα ήταν το λιγότερο αποτελεσματικό σε σχέση με το πρόγραμμα για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Τον τίτλο μας τον έχουμε διατυπώσει πρέπει να σας πω ε, με πολύ μεγάλη προσοχή και λέμε πρώιμη αξιολόγηση γιατί δεν είναι μια τελική αξιολόγηση. Πρέπει να δούμε να προχωρούν τα προγράμματα και δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε οριστικά συμπεράσματα ακόμη. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να αντιληφθούμε όταν μιλούμε για προγράμματα χρηματοδοτική ενίσχυση υποστήριξη στην Ευρωζώνη είναι ότι υπάρχει μια πολύ ιδιάζουσα δομή και εικόνα. Έχουμε να κάνουμε πολύ συγκεκριμένου περιορισμού που καθιστούν τη χρηματοδότηση στην Ευρωζώνη μέρο τη χρηματοδότηση σε σχέση με την συνήθεια χρηματοδότηση του Δουνουτού Έχουμε περιορισμούς δηλαδή και λόγω της Ευρωζώνης αλλά και της ε, ενοποίησης που υπάρχει στην Ευρωζώνη. Έχουμε προβλήματα διότι δεν υπήρχε ευρωπαϊκός θεσμός για τη χρηματοδότηση, ιδιαίτερα για την Ελλάδα αυτό ήταν ένα πρόβλημα, δεν υπήρχε, υπήρχε μάλλον η πεποίθηση ότι δεν πρέπει καν να δοθεί μέσα στην Ευρωζώνη, σε κράτος Ευρωζώνης, χρηματοδοτική ενίσχυση. Δηλαδή νομικούς περιορισμούς αντιμετωπίσαμε και με άλλα λόγια η Ελλάδα ήταν η πρώτη που δοκιμάστηκε με, αυτό, με αυτή την εμπειρία. Έξω και ήταν πολύ δύσκολη η εμπειρία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τρόικα. Τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά δηλαδή, της υπόθεσης Ελλάδας ήταν μοναδικά, στην αρχή τουλάχιστον. Δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, κόστος και αποτελέσματος. Θα πρέπει να δούμε τι διατίθεται και τι αποτέλεσμα δίνει. Στο πρόγραμμα, στα τρία προγράμματα, τα τρία μνημόνια για τις τρεις χώρες, είχαμε μεγάλο όγκο ενίσχυση σε σχέση με, τη, με τα διεθνή δεδομένα, ιδιαίτερα για την Ελλάδα. Και βλέπετε στα δεξιά στη δεξιά, στο δεξί κομμάτι της διαφάνειας το μέγεθος ως προς το ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτους όρους των μνημονίων που έχει τα τελευταία 20 χρόνια συντάξει με χώρες, τις ενίσχυση δηλαδή σε χώρες ανά τον κόσμο, το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο και αυτό αφορά μόνο το μερίδιο που ε, αφορά το Διεθνές Ομοσπονδιακό Ταμείο. Βλέπετε λοιπόν, αν δεν διαβάζετε τα γράμματα, ότι η μεγάλη αυτή ο μεγάλος δίσκος στα δεξιά είναι η Ελλάδα και πάλι μόνο στο μερίδιο του Δούνου και σε ποσοστό ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτους όρους, σε δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, έχει το μεγαλύτερο ε, πρόγραμμα η Ελλάδα. Και ξέρετε, ο Δουνουτού μόνο το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης έχει χορηγήσει. Άρα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της χρηματοδότησης για την Ελλάδα, είναι μεγαλύτερο και σε σχέση με άλλα προγράμματα που αφορούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ συγκρίνουμε με τη Ρουμανία, Λετωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και την Ελλάδα και βλέπω το ελληνικό πρόγραμμα με ποσοστό άνω του 120% επί του ΑΕΠ της χώρας ξεπερνά κάθε άλλη ε, κάθε άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα τώρα για την Ελλάδα. Μπορούμε να πούμε, πιστεύω, πως στην αρχή του προγράμματος ήταν μεγάλες οι ανισότητες, βαθέα τα προβλήματα και θα υπενθυμίσω το μεγάλο έλλειμμα τρέχουσών συναλλαγών, το τεράστιο δημόσιο έλλειμμα, το περί πολύ περιορισμένο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση, πολύ κακή δημόσια διοίκηση, όπως συζητήθηκε και το πρωί, μεγάλες δηλαδή ανισορροπίες. Το αρχικό πρόγραμμα λοιπόν, όπως είχε σχεδιαστεί, δεν ήταν αρκετά γερό, δεν ήταν αρκετά εδρεωμένο. Από την αρχή δηλαδή φαινόταν η πιθανότητα να χρειαστούν σύντομα προσαρμογές. Δεν ήταν εδρεωμένο και ως προς την βιωσιμότητα του χρέους και επιπλέον ήταν υπερβολικά αισιόδοξο ως προς τα αποτελέσματα των εσόδων από την ιδιωτικοποίηση και των φορολογικών εσόδων που θα μπορούσαν να εισπραχθούν στα προσεχή έτη. Και τρίτον, εξ αρχής, το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη φορολογία. Αν διαβάσετε τα έγγραφα τα σχετικά με το μνημόνιο, είναι σαφές το ότι η Τρόικα άλλαξε γνώμη ως προς το τι θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα. Γιατί στην αρχή επικεντρωνόταν στα δημόσια οικονομικά, κάπου στα μισά του προγράμματος βλέπουμε μια σαφή μεταστροφή όπου λέει πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα, διοικητική μεταρρύθμιση παραδείγματι, αλλά όχι μόνο, μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας και και φορολογική μεταρρύθμιση και ε, δημοσιονομική εξυγίανση καλύτερα, δηλαδή πρέπει μια σεφή μεταστροφή ή μετακύληση του βάρου στα προγράμματα. Και ζητώντα συγγνώμη γιατί είμαι οικονομολόγο και υποχρεωτικά θα σα δώσω αριθμητικά στοιχεία, θα ήθελα να σα δώσω μια πολύ απλή σύγκριση και αφήνω στο, κατά μέρο την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, μόνο για την Ελλάδα θα μιλήσουμε στην πρώτη στήλη, τι υποθέσει που είχαν διατυπώσει τα προγράμματα στην αρχή το 2010 ότι θα πώς θα ήταν η κατάσταση το 2013 κατά τις προβλέψεις του 2010 και τι εικόνα έχουμε τώρα το 2013 το Φεβρουάριο. Σε ορισμένα σημεία τα αριθμητικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτο αποτέλεσμα, ΑΕΠ, εσωτερική ζήτηση. Και τα δύο έχουν καταρρεύσει και έχουν καταρρεύσει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσε ο Ιωσδήποτε να προβλέψει. Στην αρχή του προγράμματος υπήρχε μία πρόβλεψη πως θα συρρυκνωθεί κατά 3,5% το πραγματικό ΑΕΠ. Εν τέλει έχουμε μείωση 21%. Επίσης είχε προβλεφθεί αρχικά μείωση της εσωτερικής ζήτησης κατά 11,8%, 12 περίπου έχει 28,4% πραγματική μείωση με συνέπεια και στην απασχόληση η ανεργία. Είχε προβλεφθεί πως θα φτάσει το 13. Στην αρχή του προγράμματος προβλεπόταν ότι το 13 θα είναι 15% και τελικά έχει φτάσει το 27% για την ίδια περίοδο. Υπάρχουν όμως και καλά νέα. Περιέργως πώς. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι εκεί που είχε προβλεφθεί να φτάσει, άλλωστε το επισήμαναν και άλλοι από τους ομιλητές νωρίτερα. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα δημόσια οικονομικά έχουν εξηγιανθεί σημαντικά, έχει γίνει προσαρμογή του δημοσιονομικού ελλείμματος ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, πράγμα το οποίο βεβαίως οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Γιατί αδίποτε παρεκτροπή ως προς την εξυγίανση δεν θα ε, επέτρεπε την καταβολή των δόσεων της βοήθειας. Κάτι άλλο για τους τρέχοντες, ε, για το συζύγιο τρέχουσων ε, λογαριασμών βλέπουμε μία μικρή απόκληση μόνο από τις προβλέψεις. Το γενικό χρέος έχει αυξηθεί περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί, στο 175% αντί για το προβλεπόμενο 150%. Το 150% ε, έχει προβλεφθεί χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους. Διερωτώμεθα λοιπόν γιατί τέτοια μεγάλη απόκληση και κάναμε την ανάλυση μας για να εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο πολύ υψηλότερα τα ποσοστά του χρέους μαζί με την αναδιάρθρωση από ό,τι αρχικά έχει προβλεφθεί χωρίς αναδιάρθρωση. Τρεις λοιπόν οι τομείς που εντοπίζουμε. Πρώτον, το 2009 και στην αρχή του προγράμματος οι οι οικονομικές, δημοσιονομικές συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες από ό,τι αρχικά ήταν γνωστό, εν ολίγης. Μέσα σε ένα εξάμεινο αντελήφθη η Τρόικα, ή και λιγότερο από έξι μήνες ακόμη, αντελήφθη η Τρόικα ότι ήταν 40% υψηλότερο το ποσοστό του, 14 διορθώνει ο επί του ΑΕΠ το ποσοστό του χρέους υψηλότερο από ό,τι αρχικά είχαν προβλέψει. Πρώτον, κατέρευσε το ΑΕΠ σημαντικά και άρα το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ μοιραία αυξάνεται ραγδαία, αφού έχει τόσο πολύ μειωθεί το ΑΕΠ. Αυτό εξηγεί τη μεγάλη απόκληση ως προς το δημόσιο χρέος. Ένας τρίτος παράγων που παίξε ρόλο ήταν αναδιάρθρωση του χρέους που βοήθησε στη μείωση κατά 26,6% όπως υπολογίζουμε εμείς τουλάχιστον του χρέους. Είπα ότι ήταν αισιόδοξη η Τρόικα ως προς τη... τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση στις εκτιμήσεις της. Εδώ αυτό που βλέπουμε και θα σας παρακαλέσω να κοιτάξετε μόνο τα νούμερα για το 2015 το 2015 μας δείχνει διάφορες εκτιμήσεις της Τρόικα από διαφορετικά έγγραφά της για το πόσα δισεκατομμύρια μπορούμε να περιμένουμε να έχουν εισπραχθεί μέχρι το 2015 από ιδιωτικοποίησεις. Στην αρχή του προγράμματος, το Μάιο του 2010, προβλέπει ότι θα μπορέσει να εισπράξει 5 δισεκατομμύρια από τις ιδιωτικοποίησεις η ελληνική κυβέρνηση. Όταν επιδεινώθηκε το πρόγραμμα, η προσαρμογή είχε σαν αποτέλεσμα ιδιωτικοποιήσεις με αυξανόμενα έσοδα, με μέγιστο ποσό τον Δεκέμβριο του 2011 50 αντί για 5 δισεκατομμύρια. Τώρα έχει κάπως καμφθεί η αισιοδοξία, έχει επανέλθει στο προσκήνιο ο ρεαλισμός και έχουμε πέσει κάπου στα 6 με 7 δισεκατομμύρια προσδοκόμενα έσοδα από τις ιδιωτικοποίησεις. Δηλαδή εκεί που ξέφευγε το πρόγραμμα από, το, από την πορεία του, ε, αντί να το προσαρμόσουμε και να το εδραιώσουμε, λέγαμε ότι η ιδιωτικοποίηση θα φέρει πιο πολλά έσοδα. Μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Ελλάδα επίσης έχουν σημειωθεί, συζητήθηκαν και σήμερα. Είχαμε, όπως είπα, την αναθεώρηση των συνθήκων εκκίνησης. Είπα ότι υπήρχε και μεγαλύτερη συρρήγνωση στη ζήτηση από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί. Είπα ότι υπήρχε απογοήτευση ως προς τις επιδόσεις της εξαγωγές σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα της Τρόικα, γιατί θεωρούνταν ότι θα συνέβαλε πολύ περισσότερο το μέσο των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ και βέβαια και την ε, αύξηση της ζήτησης από ό,τι τελικά όμως απεδείχθη. Είπα ότι υπήρχαν προβλήματα πολιτικά διοικητικά στην Ελλάδα και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως η Τρόικα αρχικά στην αρχή του προγράμματος υποτίμησε την δυσκολία που θα έβρισκε μπροστά της ως προς την πραγματική υλοποίηση του προγράμματος. Και αυτό διαφέρει σημαντικά από τα όσα συνέβησαν στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία, όπου η υλοποίηση σε επίπεδο χώρας, εθνικό επίπεδο, δεν είχε πρόβλημα τόσο πολύ. Και επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει ως προς την αναδιάρθρωση του χρέους, οι οποίες βεβαίως επιβάρυναν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, γιατί διαρκώς υπονομευόταν το πρόγραμμα ως προς την αποτελεσματικότητά του και τη δυνατότητα μείωσης του χρέους της Ελλάδας. Μετά όλες οι κουβέντες για το Brexit, το να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη, ε, διάφοροι μεγάλοι πολιτικοί ή υπεύθυνοι για λήψη αποφάσεων που κάνανε τέτοιου είδους δηλώσεις επιβάρυναν, ζημίωναν διαρκώς την κατάσταση, υπονόμευαν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας και ως εκ τούτου υπονόμευαν την κατάσταση στην Ελλάδα. Ως προς τις συστάσεις είναι πολύ δύσκολο να σας πω τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά και καλύτερα. Πάντα εκ των υστέρων μπορούμε βέβαια να κάνουμε υποθέσεις, αλλά θα ήθελα εγώ να επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Καταρχάς, μια πρόορη, προ, πιο νωρί αν είχε γίνει η αναδιάρθρωση του χρέους. Όχι πολύ πρόημα, όχι από την αρχή δηλαδή, γιατί θα οδηγούσε σε κόμπες καθυστερήσεις, δισταγμούς, ε, από σταθεροποίηση της οικονομίας. Αλλά το 2011 στην αρχή του έτους, αν είχε γίνει η αναδιάρθρωση του ε, χρέους και αν είχε, θα είχε μειωθεί ακόμη περισσότερο το χρέος από ό,τι πραγματικά μειώθηκε και πάνω απ' όλα θα είχε περιορίσει και την έκθεση ολόκληρης της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνούς Νομισματικού Ταμείου σε σχέση με την Ελλάδα. Το 2011 τι κάναμε, μεγάλο κομμάτι από τις θεωτικές απαιτήσει κατά εις βάρος της Ελλάδας τις αντικαταστήσαμε από δημόσιες απαιτήσει προς την Ελλάδα. Επίσης ένα πιο ε, αποτελεσματικό και αποφασιστικό πρόγραμμα, ένα πιο ρωμαλαίο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει βελτιώσει την αξιοπιστία και τις πιθανότητες επιτυχίας του ταυτόχρονα. Εν όλο θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι ακόμη στο ευρώ η Ελλάδα και αυτό ήδη αποτελεί μεγάλο επίτευγμα, αλλά η πρόσβαση στις αγορές που είναι ο τελικός στόχος του προγράμματος απέχει πολύ ακόμη. Χρειάζονται ακόμη πολλές μεταρρυθμίσεις. Και πιστεύουμε ότι θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι ότου μπορέσει η Ελλάδα να έχει ε, να απαλλαγεί πλήρως από οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης και ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ακόμα ένα λεπτό. Αν επιτρέπετε λοιπόν θα ήθελα να σας δείξω μια τελευταία διαφάνεια για την Τρόικα. την οποία δεν είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω νωρίτερα, αλλά βέβαια στην ιστοσελίδα μας, ε, στο νηστό τοπό μας είναι διαθέσιμη η έκθεση αυτή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις που αφορούν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά εν γέννη τη λειτουργία της Τρόικα. Καταρχάς θα πρέπει να παραμείνει το Διεθνές Ταμείο στο σύστημα της Τρόικα και θα πρέπει, πιστεύουμε, να αλλάξει σε μια από τις τρεις επιλογές που παρουσιάζουμε εδώ πιστεύουμε ότι η τρίτη θα ήταν η προτιμότερη ως προς το ρόλο του Διεθνούς Ταμείου, δηλαδή να είναι καταλυτικός καταλυτικής φύσεως δανειστής, να είναι δανειστής μεν, αλλά όχι ε, ο μεγαλύτερος, ένα 10% θα λέγαμε θα ήταν μια καλή συμβαστική λύση για τη συμμετοχή στο δανεισμό του Διεθνούς Ταμείου, ώστε να μπορεί και να διατηρεί την ανεξαρτησία του, αλλά και να είναι σε θέση να αποχωρήσει εφόσον το επιθυμεί από ένα μνημόνιο, από ένα πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί και να συμβάλλει σε αυτό, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Ο δεύτερο, η δεύτερη κατηγορία είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε μια παράδοξη κατάσταση ως μέλος της Τρόικα, διότι εν τέλει δεν δρά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Εκπροσωπεί ε, την Ευρωζώνη, αλλά όχι τους επιτρόπους. Δεν δρά δηλαδή ως συλλογικό όργανο των επιτρόπων. Αποφασίζει ο Επίτροπο των Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, αλλά δεν λαμβάνονται αποφάσει από το συλλογικό όργανο των Επιτρόπων για να χορηγήσουν τη σχετική εντολή. Και αυτό είναι το πρόβλημα, πιστεύουμε, γιατί η Επιτροπή έχει συλλογικό χαρακτήρα. Δεν είναι διαπραγματευόμενο εταίρο, δεν είναι μέρο των διαπραγματεύσεων. Άρα αυτό είναι εις βάρος τόσο της Επιτροπής όσο και της λειτουργίας του Μνημονίου, διότι έχουμε να κάνουμε με ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο λειτουργεί ως εκπρόσωπος κρατών μελών. Και αυτό αποτελεί βέβαια και γεννά πολλά προβλήματα. Επίσης στα, προγράμματα χρηματοδότησης, χρηματοδοτικής ενίσχυσης θα πρέπει να ε, λειτουργούν από έναν ε, θεσμό που θα έχει αναλάβει τεχνικό κομμάτι για την υλοποίηση και θα είναι σχετικά ανεξάρτητο σε αυτό. Μια επιλογή που θα μπορούσαμε να προτείνουμε ως εκ τούτου θα ήταν να μετατραπεί ο μηχανισμός σταθεροποίησης σε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο θα λέγαμε, ενός τύπου ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, ως κοινοτικός θεσμός, ως θεσμός της Ένωσης ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρική Τράπεζας. Θα πρέπει να υπάρχει, να πρέπει να συμμετέσχει, είναι κύριος δανειστής, αναλαμβάνει και εκτίθεται σε μεγάλους κινδύνους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ιδιαίτερα όταν θα αναλάβει και την εποπτεία, την τραπεζική εποπτεία, θα πρέπει να είναι σε θέση και να ενημερώνεται και να εκφράζει. Και να ενημερώνει και να εκφράζει όποιε ανησυχίε ενδεχομένω έχει. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι διαπραγματευόμενο εταίρο, μέρο των διαπραγματεύσεων. Διότι τότε βρίσκεται σε ε, αντίφαση, σε ασυμβατότητα με την πρωταρχική τη εντολή, πράγμα το οποίο αποτελεί πρόβλημα. Και έτσι πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνυπογράφει τι δηλώσει στο τέλο κάθε αποστολή τη Τρόικα. Μόνο η Επιτροπή και το Διεθνέ Προσματικό Ταμείο θα πρέπει να τι υπογράφουν. Και εν τέλει για τη βελτίωση της ε, λογοδοσία πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει τα προγράμματα, χωρί όμω ταυτόχρονα να λαμβάνει αποφάσει για αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι αυτό το οποίο θα, θα λαμβάνει τι αποφάσει. Θα πρέπει όμω να έχει μια λειτουργία επιτήρηση εποπτεία στα μνημόνια. Ευχαριστώ. Yeah, Ευχαριστώ, κύριε Γούλφ. Ήσασταν πολύ ακριβείς στο χρόνο μιλία σας και σας συγχαίρω και για τα αποτελέσματα αυτής της ε, μελέτης. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ο κύριος Κυλακάκης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Εγώ είμαι σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Το 2010 και 2011 <clears throat> είχα ζητήσει επιτάχυνση του προγράμματος περικοπές δαπανών και όχι αύξηση της φορολογίας. Και όταν ε, είχε προταθεί το ποσό των 50 εκατομμυρίων είχα πει την επόμενη μέρα ότι είχα κάνει ερώτηση στο Κοινοβούλιο το Ελληνικό ότι πρόκειται για ένα γελίο ποσό. Με πάση περιπτώσει, μεταξύ 2010 και 2012, το κύριο βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν κατά του προγράμματος για την πρώτη διετία. Σήμερα πρόκειται για το κόμμα της κυβέρνησης. Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε και ξεπέρασε τις προβλέψεις. Πώς κατά την άποψή σας αυτό που κάνετε έχει παίξει ένα ρόλο, έχει συνεισφέρει στα αποτελέσματα. Κύριος Χατζημαρκάκης, ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα επανέλθω σε αυτό στα σχόλιά μου στο τέλος της συνεδρίασης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Ράιχενμπαχ ότι αντικειμενικά έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αντικειμενικά, είπε ο κύριος Ράιχενμπαχ, αναφερόμενος σε μια νέα θέση του δημόσιου τομέα που είναι ο αρμόδιος για τη γενική επιτήρηση του προϋπολογισμού. Και πάλι μία θέση στο δημόσιο τομέα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι βελτίωση. Επίσης η Τρόικα άρχισε να έχει λίγο πιο θετικές εκτιμήσεις. Και η ερώτησή μου είναι γιατί λόγω του στόχου για την εσωτερική υποτίμηση είναι κάτι που πρότεινε εδώ στο Κοινοβούλιο ο κύριος Ράσμουσεν μιλώντας για την εσωτερική υποτίμηση που είχε σαν σκοπό ουσιαστικά την μείωση των τιμών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Κανείς δεν είναι κατά. Βεβαίως ε, σήμερα έχουμε ένα πλεόνασμα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό όμως προέρχεται από το ότι αυξήθηκε ο συντελεστής ΦΠΑ από 13-23, είτε διότι πραγματικά υπάρχει καλύτερη φόρο πρακτική ικανότητα των ελληνικών αρχών. Οι Έλληνες σήμερα αδυνατούν να καταναλώσουν περισσότερο. Και αυτοί που μας παρακολουθούν ζωντανά τη σημερινή μας συνεδρίαση, θα ήθελα να ακούσουν εάν σκοπεύετε να στηρίξετε τον ιδιωτικό τομέα. Με διάφορα μέτρα για την στήριξη της αγοράς, για τον περιορισμό της φορολογίας που πλήττει κάποιους τομείς και αν θεωρείτε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα είναι αρκετά. Ευχαριστώ Γιώργο. Ένας ακόμα συνάδελφος έχει ζητήσει το λόγο, η Νέσα Γιάλα Σέντερ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να μιλήσει, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Βόλφ, ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και τη μελέτη σας. Καταρχάς θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεδομένης τις εντύπωση που έχει δημιουργεί ότι υπάρχει μια τεράστια χρηματοοικονομική συνδρομή προς την Ελλάδα, όπως παρουσιάσατε εσείς και στους πίνακές σας ε, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγεται όσον αφορά την μικρή ικανότητα, αν θέλετε, εξυγχρονισμού και ανάπτυξης της χώρας ε, παρά την τόσο σημαντική βοήθεια. Ποιο είναι το πρόβλημα, πού έγκυται και ποιες είναι οι αδυναμίες ε, οι οποίες δεν επέτρεψαν να αποφέρει καρπούς όλη αυτή η χρηματοδότηση. Δεύτερον, μου φαίνεται ιδιαίτερα ανησυχητικό αυτό το οποίο μας είπατε, δηλαδή ότι όλες οι προβλέψεις και τα αποτελέσματα έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Ε, ακραίες σε κάποιες περιπτώσεις. Επειδή αναφερθήκατε στην Ελλάδα και μόνο, δεν ξέρω αν έχει συμβεί και σε άλλες χώρες αυτό ή όχι. Για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία ε, αναφερθήκατε αποκλειστικά στην Ελλάδα. Στην περίπτωση της Ισπανίας, από την οποία κατάγομαι εγώ, οι προβλέψεις και τα συμπεράσματα είχαν ε, ακραίες διαφορές μεταξύ των. Σε τι οφείλεται αυτό, ε, κακοδιαχείριση, ε, κακοί επαγγελματίες, πού έγινε το πρόβλημα, γιατί πραγματικά με ανησυχεί πολύ. Ε, δεν θέλουμε στο μέλλον να επαναληφθούν αντίστοιχες καταστάσεις. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα λύσουμε όλα αυτά. Και επίση ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ο κύριο Ράιχενμπαχ μα είπε και θέλω και να το πιστέψω γιατί ξέρω πώ δουλεύει με ιδιαίτερη πειθαρχία ότι είναι ένας χρόνος στον οποίο ο τουρισμός και οι εξαγωγές ε, θα έχουν μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα. Το ίδιο ακούγεται και για την Ισπανία για τις εξαγωγές. Στην Ισπανία εξηγείται για λόγους οι οποίοι δεν είναι και καλύτεροι επειδή έπεσαν τόσο πολύ οι ε, ε, και ε, λόγω της κρίσης μειώθηκαν και οι μισθοί, ε, είμαστε πιο ανταγωνιστικοί για τις εξαγωγές. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ισχύει το ίδιο. Εάν λοιπόν μας λέει ο κύριος Ράιχενμπαχ ότι οι εξαγωγές θα είναι ένας από τους ισχυρούς πυλώνες μαζί με τον τουρισμό για την ανάπτυξη της Ελλάδος, ενώ εσείς εδώ μας λέτε ότι οι εξαγωγικές δυνατότητες ε, ήταν μάλλον αποτυχημένες. Ε, και υπήρχε και μια κάποια αντίδραση προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια είναι η απόψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις εξαιρετικές σας ερωτήσεις. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω τουλάχιστον εν μέρη. Καταρχάς, η πρώτη ερώτηση νομίζω ότι δεν μπορώ να σας την απαντήσω, διότι ε, απαιτεί βαθιά πολιτική ανάλυση. Εγώ ως οικονομολόγος λοιπόν ε, δεν θα απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Να περάσω λοιπόν στην ερώτηση του κυρίου Χατζημαρκάκη για το κατά πόσον έχει αντικειμενικά βελτιωθεί η κατάσταση. Πρώτον, Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αντικειμενικά ότι η κατάσταση της χρηματοδότησης έχει βελτιωθεί ε, σημαντικά. Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης ήταν ε, καταστροφικές ε, πριν από ένα χρόνο, αλλά σίγουρα είναι καλύτερες φέτος από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Και εδώ μπορώ να πω ότι έχουμε μια αντικειμενική βελτίωση. Ένας λόγος βέβαια ε, που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή την βελτίωση δεν υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο από ακαδημαϊκής πλευράς να σας δώσουμε ένα και μόνο λόγο. Σίγουρα ε, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο το γεγονός ε, ότι οι συζητήσεις για το ελληνικό exit, την ελληνική έξοδο έχουν σταματήσει και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα κολοσσία σφάλματα και νομίζω ότι γι' αυτό ευθύνεται η Ευρώπη και όχι η Ελλάδα. Ήταν τεράστιο σφάλμα και είχε και ε, πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία. Αναφερθήκατε επίσης και ε, στην ε, εσωτερική υποτίμηση. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα ε, σφάλματα στην αρχή του προγράμματος ήταν ε, ε, το γεγονός ότι άρχισε να συζητάτε μια αρχική υποτίμηση. Υπάρχει ακόμα και συζήτηση σε πρόγραμμα της Τρόικας, το οποίο αναφέρεται στο 13ο και 14ο μισθό. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους διακόψουμε και αυτούς ή όχι, τότε η Τρόικα επισήμως έλεγε ότι δεν θα πρέπει να διακοπούν ο 13 ο και ο 14 ο μισθός γιατί θα υποσκάψουν τη βιωσιμότητα του χρέους. Αν δεν προσαρμόσει κάποιος τις τιμές, ε, ε, στις ποσότητες, ουσιαστικά έχουμε ανεργία. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ε, πολύ μεγάλο σφάλμα. Σίγουρα έχει αλλάξει η κατάσταση και τα πιο πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι μισθοί έχουν ε, μειωθεί ουσιαστικά ε, και το κόστος εργασίας έχει μειωθεί. Επομένως, από αυτή την πλευρά θεωρούμε ότι έχει αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι αυτό δεν έχει μεταφραστεί απολύτως σε τιμές. Μειώνεται το κόστος της παραγωγής, αλλά οι τιμές εξακολουθούν να είναι ακριβές. Το οποίο αφενός επηρεάζει την εσωτερική κατανάλωση, διότι εφόσον μειώνονται οι μισθοί, δεν υπάρχει χρήμα για κατανάλωση και αφετέρου μειώνεται η εξαγωγική μας δυνατότητα. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο και σχετίζεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της. Ε, υπάρχει ανταγωνισμός για, τους, ε, για τα ενίκια, για τις ε, υπόλοιπες αγορές και νομίζω ότι εδώ η πολιτική ανταγωνισμού θα μπορούσε να διαδραματίσει λίγο πιο σημαντικό ρόλο τι ακριβώς πρέπει να γίνει είναι δύσκολο να το πούμε και σίγουρα χρειάζονται ειδικοί όπως ο κύριος Ράιχενμπαχ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουν πραγματικά να εντοπίσουν πού ε, ε, θα πρέπει να εστιάσουμε και τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά τώρα το πλεόνασμα και την προσαρμογή, συμφωνώ ότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν έχει γίνει, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό, όπως θα επιθυμούσε κάποιος. Θα θέλαμε, για παράδειγμα, να την κάνουμε μειώνοντας ε, τις παραγωγικές δαπάνες, αυξάνοντας ε, τους φόρους οι οποίοι θα επηρεάσουν λιγότερο την ανάπτυξη και στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν έχει γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, Ζητάμε όμως και πολλά. Είναι πολύ δύσκολο να ε, βρούμε τη σωστή φορολόγηση και αυτό δεν αφορά μόνο το πλαίσιο της Ελλάδος, αφορά και άλλες οικονομίες. Η αντανακλαστική αντίδραση είναι πάντα να περικόψουμε τα πιο εύκολα. Ε, ε, έρευνα, επενδύσεις κλπ. και να αυξηθούν αυτά τα οποία είναι ευκολότερα να αυξηθούν το ΦΠΑ, φόροι εργασίας και το καθεξής. Και τι κάνουμε, μπορεί να θέλει κάποιος να έχει καλύτερο φορολογικό σύστημα. Αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες των φορολογικών αρχών να ε, μπορούν να συλλέγουν φόρους και από πιο ε, πλούσιες οικογένειες και πιο πλούσιες επιχειρήσεις. Ε, αυτό είναι πάντα ο στόχος ε, στη διαδικασία της φορολόγησης. Σίγουρα δεν είναι τέλεια τα συστήματα όπως είναι και αυτό σίγουρα μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε το, αυτό ισχύει και σε αυτή την περίπτωση. Για τον ιδιωτικό τομέα τώρα, αν βοηθά επαρκώ ο ιδιωτικό τομέα, Σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πέρσι. Αλλά εξακολουθώ να φρονώ ότι θα χρειαστεί χρόνος ε, προτού μπορέσουμε να έχουμε ένα βιώσιμο τομέα εξαγωγών, ο οποίος θα μπορεί πραγματικά να ε, βοηθήσει στην ανάπτυξη. Γιατί λέτε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο ιδιωτικό τομέα, Γιατί οι συνθήκε χρηματοδότηση είναι καλύτερε. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο και επομένω έχουν βελτιωθεί αυτά τα στοιχεία. Questions, um, gap in other countries. Uh, I, I didn't για τις υπόλοιπες χώρες. Δεν είχα χρόνο να μιλήσω για τις υπόλοιπες χώρες, αλλά σίγουρα στην Ελλάδα οι, οι προβλέψεις ήταν απόλυτα λανθασμένες σε σχέση με τις άλλες χώρες. Στην Ιρλανδία, στην αρχή της Τρόικα, ε, υλοποίησε τα όσα είχε προβλέψει περίπου στο 100%. Περίπου ήταν εφαρμογή ένα προς ένα, ελάχιστες αποκλήσεις. Ε, ε στην Πορτογαλία είναι λίγο ανάμεικτα τα ζητήματα, στην Ελλάδα όμως σίγουρα ήταν δραματικά τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τώρα τις εξαγωγές, νομίζω ότι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Ράιχεμπαχ ήταν ε, ε, πρόσφατες ενδείξεις ότι έχει βελτιωθεί η εξαγωγική δραστηριότητα. Εμείς εξετάσαμε το σύνολο της περίοδου και είδαμε και τις προβλέψεις και τα αποτελέσματα και από ό,τι βλέπουμε οι εξαγωγές δεν ε, αποφέρουν καλά αποτελέσματα και ήταν και αρκετά αποδυναμωμένες αυτό το διάστημα. Δεν υπήρχε καμία ανάκαμψη ουσιαστική στις εξαγωγές Τώρα, το κατά πόσον τώρα αυτή τη στιγμή ο τομέας του τουρισμού αρχίζει να έχει κάποια ανάπτυξη δεν ξέρω. Δεν έχω εξετάσει τα στοιχεία. Μπορεί και ναι, αλλά στη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου ε, οι εξαγωγές σίγουρα δεν είχαν καλά αποτελέσματα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βόλφ. Που κρατήσατε το χρόνο για να απαντήσετε σε τόσο δύσκολες ερωτήσεις. Ρίχνω καμιά ματιά στο ρολόι. Θα πρέπει να τελειώνουμε στις 12.30 και Θόδωρε πρέπει να κάνουμε 30 δευτερόλεπτα μόνο γιατί να ακούσουμε και τον Γιώργο. Ναι, 30 δευτερόλεπτα. Στην έκθεση της Τρόικα εμφανίζεται 3% λιγότερες πιστώσεις για τον ιδιωτικό τομέα εφέτος. Γιατί μας λέτε ότι πάνε καλύτερα. Μπορείτε να δώσετε μια απάντηση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ή ένα λεπτό. Αυτό που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι έχουν μειωθεί τα επιτόκια χρηματοδότησης. Τα επιτόκια δανεισμού. Δεν λέω πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχει βελτιωθεί έστω λίγο. Αλλά πάντως είναι βελτιωμένη η κατάσταση, οι συνθήκες δανεισμού Έστω και λίγο. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό το θέμα, δηλαδή δεν είναι το κυριότερο το επιχείρηματά μου εδώ. Ευχαριστώ κύριε Γούλφ και όλους τους ομιλητές. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Χατζημαρκάκη. Τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλ, και ευχαριστώ που ήσασταν πολύ σαφείς ότι η Τρόικα έχει κάνει διπλό λάθος, όπως είπατε, και αυτό έχει να κάνει και με την απουσία δημοκρατικής νομιμοποίησης. Το περιγράψατε κι εσείς εν μέρει ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το μηχανισμό σταθεροποίηση δεν διατυπώνονται από την Επιτροπή ως συλλογικό όργανο και σχετικά του δεν ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε να κάνουμε μια σκιώδη κυβέρνηση όπου ο καθένας κρύβεται πίσω από κάποιον άλλον. Εν τέλει δεν ξέρουμε το Δούνου του ήταν αυτό το οποίο ε, πίεσε για τη συγκεκριμένη απόφαση. Ήταν η ομάδα δράσης, η Task Force, ήταν η ε, κεντρική τράπεζα, οι τράπεζες και... Στρέφομαι προ την κυρία Γκρέσλε, γιατί ξέρετε είναι γερμανικό το θέμα. Οι Γερμανοί μήπω τελικά πίεσαν για να γίνει κάτι. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ράιχενμπαχ, ο οποίο ήρθε εδώ και μαζί μα έκανε αυτό το οποίο ζητήσατε κι εσεί. Δηλαδή να προσφέρει τη δυνατότητα της επισκόπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε με την ομάδα σας και είχατε την πρόθεση και τη διάθεση να συζητήσετε μαζί μας. Θα περίμενα να ήμασταν κάπως πιο ειλικρινείς, πιο ανοιχτοί στη συζήτηση αυτή. Εν αποτελεί μια αρχή όμως. Και γιατί είναι σημαντική. Είναι σημαντική διότι χάνουμε τον πολίτη. Δεν πιστεύει πια ο πολίτης σε αυτό το εγχείρημα το χρήμα είναι ένας σπάνιος πόρος. Και όταν δαπανούμε, και κύριε Γκρέσλε, κύριε Τόιρερ, κυρία Γιάλα Σέντερο, κύριο Σταυρακάκης, εγώ, όλοι μας κάθε χρόνο με τη διαδικασία της απαλλαγής εξετάζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, ότι μπορεί να υπάρχουν εσφάλματα, κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών αλλά λέμε ότι δεν υπάρχει επαρκή έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάνουμε κάποιε αλλαγέ. Δίνουμε εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να σταματήσει να βάζει φραγμού σε αυτά τα σφάλματα που εμφανίζονται. Και το κατάφερε και χαίρομαι ιδιαίτερω που το κάνει αυτό. Και επί παραδείγματι, κάποια κράτη όπω η Ρουμανία ήρθαν για να πούνε στι Βρυξέλλε πού είναι τα λεφτά και η, Ρουμα... Επιτροπή του είπε: Α, κοιτάξτε, σταμάτησε η ροή του χρήματο, διότι είπε έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα γίνει γιατί υπήρχαν πολλά λάθη στην εκτέλεση. Για την Ελλάδα όμω, το παράδειγμα τη Task Force δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και στην προκείμενη περίπτωση, όπως είπε και ο κύριος Ράχενμπαχ, μεγάλος όγκος πόρων δόθηκε σε ένα κράτος μέλος για να βοηθηθεί το κράτος μέλος αυτό να βγει από το χάος. Γιατί η κατάσταση, συνοχή, περιφερειακή πολιτική και ούτω καθεξής πήγαινε ατέρμονα να απορροφά χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου χωρίς να δίνει αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει χάος αστικά. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε μια χώρα να καταστεί πιο αποτελεσματική. Ο κύριος Ράχενμπαχ είπε ότι σε ένα περίπου χρόνο, έτσι δεν είπατε, σε ένα χρόνο περίπου περιμένετε αυτά τα πολύ αρνητικά στοιχεία, ποσοστό 27% στην ανεργία, 62% για τους νέους η ενεργεία και λεφτά να πέσουν τα αρνητικά αυτά στοιχεία και να αρχίσει να ανθίζει κάπως η οικονομία. Γιατί στην πραγματική οικονομία αυτό βλέπει ο άνθρωπος, αυτό βλέπει ο πολίτης, δεν μπορεί να περιμένει δηλώσεις και προθέσεις. Αυτό δεν είπατε κύριε Ράχενμπαχ. Ο κύριος Ράχενμπαχ δυστυχώς δεν έχει μικρόφωνο να μένω. Διαρθρωτική αλλαγή. 32 μήνες. 32 μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε η δουλειά της ομάδας δράσης, της Task Force. Και γι' αυτό αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως ό,τι κάνουμε εδώ το κάνουμε εκ μέρου του Ευρωπαίου πολίτη και η ομάδα δράσης και ίσως θα πρέπει στο εγγύης μέλλον πάλι να την ε, έχουμε κοντά μας και θα πρέπει να ε, ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό ουσιαστικό ανταλλαγή γνώσεων, όχι μόνο θέσεις εργασίας, όχι μόνο δημοσιεύσεις ε, εκθέσεων αλλά ουσιαστικά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία και για τους Έλληνες ιδιαίτερως, γιατί και οι Έλληνες Ευρωπαίοι είναι και ως πραγματικός Ευρωπαίος και εγώ στο πλευρό των, Ευρω... των Ελλήνων είμαι και σας ευχαριστώ πολύ και τη Γραμματεία ιδιαίτερως που μας βοήθησε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση γιατί τα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζημαρκάκη. Ξέρουμε ότι είστε πάντα πολύ δραστήριος ως εισηγητής Ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν το λόγο. Εγώ ως, εισηγητής, ως πρόεδρος συγγνώμη, της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, τον κύριο Χόρστ Ράικενμπαχ, τον κύριο Στέφανο Μάνο, τον ε, κύριο Νόρμουν Σπόπεν, τον κύριο Πέτερ Στουπ Γιόργενσεν, τον κύριο Μπεν Κνάπεν, τον κύριο Γκούντραμ Βόλφ και βέβαια τον κύριο Γιώργο Χατζημαρκάκη, ο οποίο έκανε την προετοιμασία αυτή τη συνεδρίασης. Είμαστε η Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού θέτουμε τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων πολύ σοβαρών προβλημάτων. Από την άλλη εντοπίζουμε και το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο όπως έχει χρειάζεται και θα μπορούσε και να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει. Ευρωπαϊκά κονδύλια δαπανώνται στην Ελλάδα χωρίς ακόμη να υπάρχει δυνατότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να παρεμβαίνουμε. Και κλείνω με τα λόγια του κυρίου Βόλφ ότι ο στόχος του δημοσιονομικού ελλείμματος, αντιμετώπιση του μεσονομικού ελλείμματος έχει επιτευχθεί. Επιτεύχθη λοιπόν ο στόχος του μηδενισμού του ελλείμματος, αλλά με συνέπειες σοβαρές στην πραγματική οικονομία και άλλους τομείς. Άρα πρέπει τώρα να διερωτηθούμε και εμείς όπως και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και στους λοιπούς τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κάποια άλλη στιγμή. Διακόπτω προς το παρόν τη συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.